Καλημέρα σε όλους. Βλέπω πως οι δύο συνεισηγητές για το επόμενο θέμα είναι ήδη εδώ και τους καλωσορίζω θερμά. Επίσης να καλωσορίσω την ομάδα από την DG ταξού τον κύριο Ζελίνσκι, που είναι πολύ γνωστό σε όλους μας για την εργασία του όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των τελωνίων και καλωσορίζω και την, και την κυρία Άννα Γουλή που θα κάνει μια παρουσίαση για την πρόταση αυτή. Κάποιες ανακοινώσεις για να σας θυμίσω πως αυτή η συνεδρία συνεδρίαση μεταδίδεται στο ίντερνετ και επίσης ε, ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε λίγο αργότερα. Να σας θυμίσω ότι συμφωνήσαμε να αλλάξουμε τη σειρά, οπότε να ψηφίσουμε πρώτα δηλαδή την ε, πρώτη πρώτα την έκθεσή του μάλλον. Οπότε, τώρα, ε, σε λίγο θα ακούσουμε για την Κομισιόν. Πρόκειται για μια νέα πρόταση για την παραβίαση των ε, τελωνίων και σχετικής κυρώσεις. Δεν θα έχουμε τον χρόνο να το εξετάσουμε σε αυτή τη θητεία, αλλά έχει ήδη δουλέψει πάνω σε αυτό το θέμα η Επιτροπή μας μαζί με την εισηγήτρια για το πακέτο των ε, τελωνίων και έτσι ε, θέλαμε να έχουμε μια εικόνα για την πρόταση ε, και να κάνουμε και κάποιες πολιτικής φύσης παρατηρήσεις υπό τη μορφή ενός ψηφίσματος. Επίσης, επειδή είναι ένα κοινό σχέδιο, προκαλέσαμε το ΕΛΚ και τους σοσιαλιστές να ορίσουν συνεισηγητές. Η κυρία Κέπχαρντ ανέλαβε από ε, του σοσιαλιστές και η κυρία Ντερούπ από το ε, ΕΛΚ. Θα καλέσω λοιπόν τις συνεισηγητρίες να, κάνουν, να σχολιάσουν, καθώς και τους συναδέλφους που μπορεί να παρακολουθούν το θέμα και θα συμβάλλουν και στο ψήφισμα. Και έπειτα έχουμε μία πρόταση για χρονοδιάγραμμα από τις συνεισηγήτριες. Θα σας τη δώσω στο τέλος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια ένα σχετικό ψήφισμα πριν ε, τελειώσει η θετία μας. Η κυρία Αναμπολή νομίζω θα μιλήσει πρώτα και ίσως και ο κύριος Ζελίνσκι να θέλει να κάνει κάποια εισήγηση. Μετά θα σας δώσω το λόγο για ερωτήσεις. Thank you very much, Mr. Chairman. Just a very short, uh, very short introduction. And first I have to say... Μια σύντομη εισήγηση. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πολύ εσάς, την κυρία Λεγκρίπ, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για όλη την προσπάθεια που έχει γίνει για τον τελωνιακό κώδικα. Πρέπει να το πω, παρότι δεν είναι στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Έπρεπε να το αναφέρω. Έπειτα, για την ε, παρουσίαση αυτή που θα σας κάνουμε, είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα, μια πρωτοβουλία της ταξού των συναδέλφων, ε, φίλων και συνεργατών και ελπίζω ότι θα το αντιληφθείτε ότι όντως πρόκειται για μια μεγάλη προσπάθεια, μεγάλο εγχείρημα. Είναι ένας από τους ακρογωνίους λήθου ένα από τα στηρίγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δείτε πώς διαφέρει η κατάσταση στα κράτη-μέλη και είναι ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα ώστε να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Αναμπόλευ, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα σας κάνω μια σύντομη εισήγηση για το τι προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί τη βάση της εναρμόνισης όσον αφορά τις παραβιάσεις του ελληνικού κώδικα και τις σχετικές κυρώσεις. Καταρχήν να σας πω πώς προέκυψε αυτή η ιδέα. Πολλές φορές ακούσαμε στο παρελθόν ε, το Κοινοβούλιο να λέει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι όσον αφορά την διαφορά για τα εσωτερικά ε, τις εσωτερικές ρυθμίσεις των κρατών μελών για την παραβίαση των τελωνιακών κανονισμών. Ε, θέλαμε λοιπόν να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει στα κρατημέλη και ξεκινήσαμε το 2008 μέσω του Customs 2013 εκπονώντας ένα πρόγραμμα με 24 κατημέλη που εθελοντικά συμμετείχαν ώστε να διαπιστώσουμε ποια ήταν η κατάσταση σε σχέση με τις ε, παραβάσεις και τις κυρώσεις. Τα συστήματα διέφεραν κατά πολύ και θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ παράξενο να έχουμε ε, μια απόλυτα εναρμονισμένη ε, νομοθεσία, δηλαδή ε, τον τελωνιακό κώδικα και ε, μετά στη συνέχεια να έχουμε διαφορετικούς τρόπους επιβολής αυτής της συναρμονισμένης κατά άλλα νομοθεσίας. Είδαμε λοιπόν γενικά την βασική έκθεση του 2010, εργαστήκαμε επί δύο χρόνια με τα 24 κράτη εθελοντές και η έκθεση αυτή μας έδειξε ότι 16 από τα 24 κράτη μέλη έχουν ένα μεικτό σύστημα για ποινικέ και μη ποινικέ κυρώσει όσον αφορά τι παραβιάσει των τελωνίων. 8 από τα 24 κράτη-μέλη ε, προέβλεπαν μόνο ποινικέ κυρώσει, που σημαίνει ότι ακόμα και για μικρέ παραβάσει έπρεπε να περάσει κανείς από το ποινικό δίκαιο. Έπειτα, σε αυτή την κατηγορία των 8 κρατών μελών που προέβλεπαν ποινικέ κυρώσει, είχαμε ε, και ε, οικονομικά κατόφλια που αποτελούσαν το όριο ανάμεσα στο ποινικό και μη ποινικό δίκαιο. Και αυτό το κατόφλι ήταν ανάμεσα στα 216 ευρώ και τις 50 66 ευρώ και τις 50.000 ευρώ. Επίσης είχαμε αυτό που αποκαλείται αυστηρή ευθύνη παράβασης. Εδώ θεωρείται, θεωρείται στεκμήριο η παραβίαση Βλέπετε λοιπόν μια μεγάλη ποικιλία ε, κυρώσεων και θεωρήσαμε πως αυτό είναι παράξενο στην ε, Τελωνιακή Ένωση και την εσωτερική αγορά όπου έχουμε οικονομικούς φορείς οι οποίοι χρειάζεται να εργάζονται σε ισότιμη βάση και επίσης στο τελωνιακό κώδικα, όπως γνωρίζετε, έχουμε προβλέψει την έννοια του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, όπου ε, η πρόσβαση σημαίνει την πλήρωση διάφορων κριτηρίων. Ένα εξ αυτών είναι η συμμόρφωση προς την τελωνιακή νομοθεσία. Φαντάζεστε ότι, ότι αν συμμορφούνται κανείς προς ένα προς την νομοθεσία όπου δεν προβλέπεται ας πούμε, σε κάποιο κράτος μέλος ε, ποινή ενώ σε κάποιο άλλο μέλος ε, προβλέπεται ποινή για συγκεκριμένη παράβαση ποινικού χαρακτήρα ε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ισότιμο πεδίο. Επίσης και έχουμε διαφορετικά χρονικά όρια στα κράτη-μέλη όσον αφορά τις κυρώσεις από το 1 έως το 30 έτη. Επίσης κάποια κράτη-μέλη δεν προβλέπουν κανένα απολύτως χρονικό όριο. Φαντάζεστε λοιπόν ότι σε έναν, σε έναν ε, κόσμο επιχειρήσεων όπου είσαι οικονομικός φορέας και αναμένεις απόφαση για να εκτιμήσεις αν είσαι ένοχος για μια παράβαση ή όχι, μπορεί να περιμένεις και για πάντα. Μπορεί να πτωχεύσεις εντωμεταξύ και θεωρήσαμε ότι και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Διαφορετική κατάσταση ισχύει και για την ευθύνη των διαφόρων ε, νομικών προσώπων, γιατί στα 15 κρατημέλη από τα 24 υπήρχε η ευθύνη για το νομικό πρόσωπο, ενώ, πρόσωπο, ενώ στα υπόλοιπα όχι. Αυτό είναι προβληματικό όχι μόνο εν γέννη για το δίκαιο, αλλά και για το κόστος του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Έχουμε επίση κάποιε κυρώσει που ονομάζονται ε, ρυθμίσεις, στα διακανονισμοί μάλλον, στα κράτη-μέλη. Δηλαδή υπάρχει κάποια ποινή που προβλέπεται από τον νόμο, αλλά, προσπαθώ να βρω ένα διακανονισμό ανάμεσα στη διοίκηση, τα τελωνία και τον οικονομικό φορέα για να βρεθεί μια συμφωνία όσον αφορά την ποινή. Είναι μια αδιαφανή διαδικασία και τα 15 από τα 24 κράτη-μέλη είχαν τέτοιου είδου διαδικασία. Τα κράτη-μέλη που προβλέπουν αυτού του είδου του διακανονισμούς είναι αυτά που ε, προβλέπουν μόνο ποινικού τύπου κυρώσει για τις παραβιάσει των τελωνίων. Φανταστείτε την εξή κατάσταση. Μια εταιρεία ξεκινά μια δήλωση εξαγωγή στο τελωνιακό γραφείο δύο μέρες ε, μετά από τη φόρτωση των αγαθών στο εμπορευματοκιβώτιο. Εδώ υπάρχει παράβαση. Σε ένα κράτος μέλος δεν θεωρείται παράβαση καθόλου οπότε δεν προβλέπεται κύρωση. Σε νέα κρατημέλη, εδώ πρόκειται για ποινική παράβαση και υπάρχουν δύο είδη ποινής, χρηματική, που μπορεί να είναι ποινικού τύπου, από 1.250 ευρώ μέχρι και 1.800.000 ευρώ. Αυτά είναι τα στοιχεία του 2010. Το ποσό ίσως να έχει αλλάξει μεταξύ, αλλά βλέπετε πόσο τεράστια είναι η διαφορά ακόμα και εντός του ίδιου είδους ε, ε, ποινής. Δύο από τα κράτη-μέλη που προβλέπουν ποινικέ παραβάσεις προβλέπουν και φυλάκιση για αυτού του είδους την κατάσταση. Μη ποινικέ κυρώσει σε 15 κράτη-μέλη που προβλέπουν οικονομικά πρόστιμα από 393 ευρώ μέχρι τα 500.000 ευρώ και 15 κράτη-μέλη τόσο σε ποινικό ή μη ποινικό δίκαιο προβλέπουν τη διαδικασία διακανονισμού. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο κράτη που δεν θεωρούν καθόλου παράβαση αυτή την κατάσταση και το κράτος μέλος που επιβάλλει ποινική φύσης πρόστιμο της τάξης του 1.800.000 εκατομμυρίου 800.000 ευρώ και ακόμα και ποινή ε, ε, φυλάκισης. Of course, this proposal has been uh, has been uh, drafted, uh, not being on an island, on a customs island. Ε, λοιπόν, ε, αυτή την πρόταση την έχουμε υποβάλει γιατί ξέρουμε ότι όλες αυτές οι ε, μάλλον οι διάφορες προτάσεις επηρεάζουν τις παραβάσεις τις τελωνιακές. Δεν ζούμε απομονωμένοι μέσα σε ένα τελωνιακό κόσμο επηρεάζονται ας πούμε από την ε, πρόταση ειδική για την καταπολέμηση των απατών ε, έναντι των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ούτω καθεξής. Και προσπαθήσαμε να συντονίσουμε τα μέσα με τα άλλα υπάρχοντα ε, μέσα ή προτάσεις. Υπάρχει και ο κανονισμός του Συμβουλίου του 95 για το ίδιο θέμα που αφορά τις μη ποινικές και φυσικά λάβουμε υπόψη τον ε, τελωνιακό κώδικα που πια σας είναι πολυκείος και βασίσαμε μάλιστα την πρότασή μας, τουλάχιστον τον κατάλογο των παραβάσεων, ε, αποκλειστικώς στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον τελωνιακό κώδικα της Ένωσης. Just a few words on the, on the relationship between the... Δύο λόγια για την σχέση με την ε, οδηγία PIF, όπως λέγεται. Κομμάτι του παιδιοφαρμογής είναι κοινό, αλλά όχι, δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση. Αυτό που ταυτίζεται είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων και έχουμε και εμείς ένα κομμάτι της οδηγίας μας που σχετίζεται με τα τελωνιακά τέλη. Αλλά όπως γνωρίζετε πρόκειται για προστασία όχι μόνο των εισοδημάτων αλλά και προστασία της κοινωνίας από απειλές στην ασφάλεια και εξασφαλίζει πως όλες ε, οι τυπικές διαδικασίες πληρούνται ακόμα και αν δεν ε, διακυβεύονται τελωνιακά τέλη. Εν μέρη λοιπόν είναι κοινό το πεδίο εφαρμογής. Τώρα, εκεί όπου έχουμε κοινό πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να αποφύγουμε την επανάληψη, ε, την επικάλυψη. Να βρούμε δηλαδή συγκεκριμένα κριτήρια όπου αυτή η οδηγία ισχύει και όπου, και η μελλοντική οδηγία PIF θα ισχύσει. Ας πούμε, στην PIF υπάρχει ένα κατόφλι 10.000 ευρώ όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα. Επίσης υπάρχει ο αποκλεισμός ε, χωρίς πρόθεση. Είναι, και εμείς στην οδηγία μας έχουμε αυτό που ονομάζουμε ε, αυστηρή παράβαση ευθύνης. Ε, θεωρούμε δηλαδή πως η πρότασή μας είναι συμπληρωματική στην οδηγία PIF και σε κάθε οδηγία που προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα ε, της Ένωσης. Και τέλος, έχουμε και έναν ε, άρθρο στον Τελωνιακό Κώδικα που ε, προβλέπει ποινές. Πριν να σας πω ακριβώς περί τίνος πρόκειται στην οδηγία, θα σας πω γιατί πιστεύουμε πως η οδηγία, η διασυνοριακή για τις παρα... τελωνιακές παραβάσεις είναι πολύ σημαντική, γιατί σήμερα οι δουλειές ε, ε, ενός οικονομικού φορέα στην Ένωση δεν είναι μόνο ευρωπαϊκού τύπου, αλλά μπορεί να είναι και παγκόσμια. Δηλαδή, ε, ε, κάποιος οικονομικός φορέας που έχει παρεδώσει ε, είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να εντοπίσει κανείς πού έγινε η παράβαση και πώς θα την ε, καλύψει. Χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στις τελωνιακές αρχές, χρειάζεται να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, την ε, παράβαση του νόμου. Αλλά δεν έχουμε μια κοινή οδηγία, δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε το διασυνοριακό στοιχείο αυτής της κατάστασης. Γι' αυτό και θεωρήσαμε πως υπάρχει ανάγκη για κοινή αναφορά και ήταν προφανής αυτή η ανάγκη. Ε, επίσης έχουμε άλλες πολιτικές που ας πούμε ε, ε, ε, η γεωργική πολιτική, ο ΦΠΑ κτλ. που δίνουν σε όλους αυτούς τους πελάτες έναν βασικό κεντρικό ρόλο και αυτό σημαίνει όχι μόνο συνεργασία ανάμεσα στις θελωνιακές αρχές αλλά και συνεργασία ανάμεσα στις θελωνιακές αρχές και άλλες αρχές άλλων κρατών μελών. Και φυσικά λάβαμε υπόψη στην περίπτωση των διασυνοριακών συναλλαγών την αρχή το ότι ε, δεν μπορούμε να ε, και δεν χρειάζεται να τιμωρείται ο παραβάτης δύο φορές ή διπλά. Ας δούμε τώρα ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της πρότασής μας, ποιος είναι ο στόχος μας σας το θυμίζω εν συντομία, είναι να γεφυρώσουμε τα κενά ανάμεσα στα διάφορα νομικά καθεστώτα που σας εξήγησα πριν για να έχουμε πιο ομοιόμορφη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Τελωνιακού Δικαίου σε όλη την επικράτεια της Ένωσης μέσω ενός κοινού καταλόγου παραβάσεων, μια κοινή ονοματολογία συμπεριφορών που αποτελούν παραβίαση του τελωνιακή της νομοθεσίας και αυτό είναι το τμήμα της εναρμόνισης, οι παραβάσεις. Έχουμε και ένα τμήμα το οποίο δεν είναι απόλυτα εναρμονισμένο, διότι θεωρήσαμε από την μελέτη των 24 κρατών μελών πως δεν ήταν δυνατόν να εναρμονίσουμε τα εθνικά νομικά καθεστώτα. Θα σήμαινε αυτό μεγάλη ε, επανάσταση. Πολιτικός θα ήταν ε, αυτοκτονικό γιατί τα κράτη-μέλη ε, επιθυμούν να διατηρήσουν τα νομικά του συστήματα πάνω κάτω. Ωστόσο, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να καλυφθεί το κενό μέσω της παροχής μιας κοινή πλατφόρμας ποινών. Ένα κοινό πλαίσιο λοιπόν για την επιβολή των ποινών σε σχέση με το τι είδους ποινές ε, επιβάλλονται και ποια είναι η κλίμακα των κυρώσεων εντός των οποίων υπάρχει μια κάποια ευελιξία. Το νομικό εργαλείο που επιλέξαμε για να διατηρηθεί αυτή η ευελιξία ήταν η οδηγία. Μπορούσαμε να είχαμε προτείνει κανονισμό, αλλά θεωρήσαμε πως έπρεπε να ε, σεβαστούμε τις διαφορές στην νομική ε, δομή και να αφήσουμε και κάποιο περιθώριο στα κρατημέλη για να μεταγράψουν αυτά τα νέα στοιχεία στην εθνική τους νομοθεσία. Γι' αυτό και επιλέξαμε την οδηγία τελικά. Ε, έτσι λοιπόν θεσπίσαμε έναν κοινό κανόνα, ε, ένα κοινό κατάλογο παραβάσεων που βασίζεται απόλυτα και αποκλειστικά στον τελωνιακό κώδικα. Αν δείτε την περιγραφή των παραβάσεων θα δείτε και την αναφορά στα διάφορα άρθρα στον τελωνιακό, του τελωνιακού κώδικα. Έχουμε τρεις κατηγορίες λοιπόν παραβάσεων, την αντικειμενική ευθύνη που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αναζητηθεί η ενοχή, η πρόθεση, οποιοδήποτε υποκειμενικό στοιχείο. Αυτές είναι ίσονος σημασίας παραβάσεις που είναι βασικά τυπικές παραβάσεις γιατί καταλάβαμε ότι κάποια καρτιμάλη έχουν πρόβλημα όσον αφορά την ε, παράβαση αυτού του τύπου αντικειμενικής ευθύνης. και έπειτα έχουμε ε, τις ε, παραβάσεις εξαμελίας και τις ε, εκπροθέσεως παραβάσεις που όπως μπορείτε να φανταστείτε ξεκινάμε από τις λιγότερο σημαντικές, πάμε στις μεσές που έχουν γίνει λόγω αμέλειας και έπειτα είναι πολύ πιο σοβαρό όταν έχουν γίνει εκπροθέσεως. Για κάθε είδος ε, παράβαση που σας ανέφερα, ε, για κάθε κατηγορία έχουμε μια κλίμακα κυρώσεων ε, και επινών που να είναι αναλογικές και αποτρεπτικές. Επιλέξαμε τις οικονομικές κυρώσεις γιατί διαπιστώσαμε πως αυτό ήταν το κοινό στοιχείο στα 24 κράτη-μέλη τα οποία συνέβαλαν ενεργά σε αυτή την έκθεση του 2010 είτε πρόκειται για ποινικού τύπου είτε όχι ε, κυρώσεις, όλα τα κράτη-μέλη, όλες οι κατηγορίες κρατών μελών έχουν ε, προβλέψει οικονομικές κυρώσεις, χρηματικά πρόστιμα δηλαδή, και τα κριτήρια που επιλέξαμε, ε, και αυτή ήταν μεγάλη μας ανησυχία, δεν ήταν ε, η αποφυγή του τελωνιακού τέλους, αλλά η αξία το τέλους ή ένα συγκεκριμένο ποσό σε περίπτωση όπου δεν ε, προβλέπονταν τελωνιακοί δασμοί. Βέβαια, ε, στα κράτη-μέλη έχουμε τους επιβαρυντικούς παράγοντες ε, είτε τα ελαφρυντικά στοιχεία για να δούμε αν αυτό το, το, το κάθε θέμα Ε, μπορεί εδώ δηλαδή να λάβουμε υπόψη διάφορες περιστάσεις σε κάθε κράτος μέλος αν όντως ισχύουν διάφορα ελαφρυντικά ή επιβαρυντικά στοιχεία. Έχουμε καθιερώσει την ευθύνη των νομικών προσώπων και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καθιερωθούν κάποιοι κανόνε για την ευθύνη των νομικών προσώπων. Αυτό δεν είναι τίποτα καινούριο, γιατί στην οδηγία ΠΙΦ υπάρχει ένα σχετικό άρθρο για την ευθύνη των νομικών προσώπων. Ορισμένε δικονομικέ πτυχέ δεν θέλαμε να μπούμε στι ε, λεπτομέρειε τη διαδικασία λόγω ακριβώς της ευελιξίας και λόγω του σεβασμού που έχουμε για τις ε, διαφορές των ενωμών τάξεων. Παρ' όλα αυτά είχαμε την αίσθηση ότι θα έπρεπε να κάνουμε κάτι για την περίοδο περιορισμού των διαδικασιών όσον αφορά τις τελωνιακές παραβάσεις και αυτό θα το βρείτε στο άρθρο 13. Θα πρέπει να ανασταλούν οι διαδικασίες όπου υπάρχουν παράλληλες ποινικέ ε, διαδικασίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει εναντίον του ιδίου προσώπου σε σχέση με τα ίδια περιστατικά και το και εφόσον πρόκειται για τα ίδια περιστατικά, θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση είτε στο πλαίσιο μια ποινική διαδικασία, ε, μελλοντικά μάλλον θα επάγεται στην ε, οδηγία PIF, είτε όχι. Αλλά ορισμένε φορέ δεν υπάρχει ο ίδιο τύπο χαρακτηρισμού, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια διασύνδεση με αυτή την παραβίαση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ανασταλεί η διαδικασία και θα πρέπει να αναμένουμε το αποτέλεσμα τη ποινική διαδικασία. Και επίση έχουμε προβλέψει ε, ποιο είναι το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση της παραβίας σε περίπτωση που ενέχονται περισσότερα από ένα κράτη. Και το θέμα της ε, εδαφικής αρκαιρεότητας, γιατί το διασυνερικό στοιχείο είναι ιδιαίτερο σημαντικό σε αυτό το πεδίο. Έχουμε προβλέψει ένα άρθρο για τη συνεργασία μεταξύ τελωνιακών αρχών, λόγω ακριβώς του ισορυνικού στοιχείου και επίσης μέχρι τη στιγμή που θα εφαρμόσετε τις ε, ουσιαστικές ε, κυρώσεις για τελειωνιακές παραβιάσεις θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα προσωρινό μέτρο του ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορείτε να πάρετε κάτι από το δράστη. Ε, άρα λοιπόν έχουμε ένα σχετικό άρθρο που προβλέπει μια κατάσχεση των αγαθών στην περίοδο αναμονής, ε, κατάσχεση των εργαλείων ή μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για να διαπραχθεί η παράβαση. Αυτό, αυτή δεν είναι σημαντική κύρωση, γιατί σαν ε, κύρωση αυτή καθ' αυτή ε, εξισώνεται με μια μορφή κατάσχεση που ήδη υπάρχει σε ορισμένε χώρε μέλη. Εν κατακλείδη λοιπόν, θεωρήσαμε ότι παρόλο που κατά πάσα πιθανότητα στα μάτια του Κοινοβουλίου ε, δεν θεωρείται ιδιαίτερος θαραλέα η πρόταση αυτή. Έπρεπε να επιλέξουμε να είμαστε πραγματιστές, ρεαλιστές. Ε, και, δεν λέω, δεν, ότι δεν υπήρξαμε ιδιαίτερα θαραλέα, δεν προτείναμε μια απόλυτη εναρμόνιση. Παρ' όλα αυτά έχουμε την αίσθηση ότι η πρόταση είναι εξορροπημένη και πραγματικά λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των χωρών μελών. Βασίζεται σε κοινά χαρακτηριστικά έτσι όπως έχουν αναγνωριστεί στη βάση της έκθεσης των χωρών μελών το 2010. Βεβαίως επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεων με τα δύο θεσμικά όργανα, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Και τέλος θα ήθελα να παραπέμψω στον Αναξίμαντρο, ο οποίος είπε ήταν ένας Έλληνας φιλόσοφος από τη Μίλητο και λέει αναφέρεται στη γένεση και η γένεση οδηγεί στη φθορά κατά το χρέον ε, για την απόδοση της δίκης ε, σύμφωνα με την αξιολόγηση του χρόνου. Γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί ορισμένοι από εξχωρισμένοι μας είπαν ότι έχετε προσπαθήσει κατ' επανάληψη από τη δεκαετία του 80 να αναγνωρίσετε τις κυρώσεις. Γιατί θέλετε να το κάνετε τώρα, γιατί η απάντηση γιατί έχουμε την αίσθηση ότι τώρα ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, γιατί τώρα υπάρχει μια σφαιρικότητα και τώρα θα πρέπει να γίνει κάτι για τους ε, οικονομικούς ε, παρόχους και να καλύψουμε τα κενά για τις διάφορες μορφές ε, ποινικών παραπτωμάτων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ξεκάθαρη παρουσίασή σας και είναι πολύ καλό κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας που παραθέσετε το απόσπασμα του Έλληνα φιλοσόφου. Ε, θα ήθελα να μας συγχωρέσετε για την ιδιαίτερα ρεαλιστική προσέγγιση, αλλά αυτή είναι μια βρετανική ε, προσέγγιση, αλλά αυτή η Επιτροπή, Επιτροπή συγγνώμη, θέλει να σημειώσει κάποιες υλικές ε, πραγματικές πρόοδους όσον αφορά τα θέματα. Νομίζω ότι τα μέλη θα έχουν αντίγραφα από την μελέτη αντιχτύπου και μια σύνοψη σε διαφορετική μορφή από τις προηγούμενες αξιολόγεις, αξιολογήσεις, συγγνώμη, αλλά είναι πολύ χρήσιμη. Τώρα, ας ακούσουμε τι σκέφτονται οι συνάδελφοι που έχουν εργαστεί σε αυτό το τομέα. Η κυρία η κυρία Λεγκρίπε, η κυρία Κέπχαρτ και οποιοδήποτε άλλος θέλει να σχολιάσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να καλημερίσω τους συναδέλφους και βέβαια να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σαφέστατη, πολύ συγκεκριμένη αυτή παρουσίαση που την ε, διαπνέει αυτός ο ρεαλισμός ε, που αναφέρατε και στο τέλος της ομιλίας σας και επίσης παιδαγωγική με επιχειρήματα. Μου άρεσε και μένα η αναφορά στην ε, αρχαιοελληνική φιλοσοφία που κάνετε στο τέλος της παρουσίασής σας στους σημερινούς καιρούς η αναφορά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ότι δεν ξεχνάμε ότι εδώ είμαστε και για κάποιες ιδέες, κάποιες ιδέες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη. Δεν είναι κάτι περιττό. Ε, απριόρι είμαι θετική σε αυτό το σχέδιο οδηγίας. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι και με ένα βλέμμα προσεκτικό αλλά θετικά διακείμενο ε, βλέπω αυτή την ε, οδηγία και με ενδιαφέρον. Αυτό το σχέδιο οδηγίας, κατά την άποψή μου, εντάσσεται σε μία συνέχεια του έργου που ξεκίνησε στην ε, παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων για τον εξυγχρονισμό, την προσαρμογή ε, την ε, περαιτέρω επεξεργασία αυτού του τελωνιακού κώδικα. Ξέρουμε όλοι ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος που έχουμε στη θέση μας και αν θέλουμε να προχωρήσουμε και να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου δεν έχουμε παραλαμβάνω πολύ χρόνο γι' αυτό και χρειάστηκε να κάνουμε μια επιλογή τακτική και στρατηγική θα τη χαρακτήριζα και μιλώ για μας τα μέλη της Επιτροπής ΙΜΚΟ πώς δηλαδή θα έπρεπε να χειριστούμε την ε, δουλειά μας ακριβώς. Και η επιλογή που κάναμε ήταν να προχωρήσουμε με ένα ψήφισμα και όχι με ένα έγγραφο εργασίας. Θεωρήσαμε ότι αυτή είναι η λύση και αυτό είναι το πιο κατάλληλο εργαλείο. Με τη συνάδελφό μου και συνεισηγήτρια Εύελιν Γκέπχαρτ από την Επιτροπή ΙΜΚΟ θελήσαμε, αν βέβαια προχωρήσουν οι εργασίες μας, να ε, Υποβάλλουμε ένα ψήφισμα δυνάμει το άρθρο 110 εδάφιο 2 του εσωτερικού μας κανονισμού ελπίζω παραλαμβάνω πριν το τέλος αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Τι σημαίνει κατάθεση ψηφίσματος. Επειδή είναι πολύ ε, σύντομα τα χρονοδιαγράμματα δεν θα μπορέσουμε βέβαια να μπούμε σε λεπτομέρειες και να τελειοποιήσουμε τις παρεμβάσεις και τη συνεισφορά μας. Απλά θέλουμε να έχουμε έτσι μια συνολική σφαιρική προσέγγιση και τοποθέτηση για τη σκοπιμότητα και τη σημασία αυτού του σχεδίου οδηγίας. Επαναλαμβάνω ότι κατά την άποψή μας πρέπει να αντικατοπτριστεί όλη η δουλειά που έχουμε κάνει στα τελωνιακά θέματα σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, δίνοντας έμφαση στον τελωνιακό κώδικα της Τελωνιακής Ένωσης. Και ελπίζω αυτό το ψήφισμα που θα σε ο Πέρας ε, να αντικατοπτρίζει και τη δική μας θέση, τη φιλοσοφία μας, αν θέλετε, για τα πλεονεκτήματα της ε, Τελωνιακής Ένωσης ε, και τον τρόπο με τον οποίο ενισχύεται και παγιώνεται. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω, όπως έκανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το παράδοξο των τελωνιακών διατάξεων. Είναι κάτι βέβαια επίκαιρο, το βλέπουμε κάθε μέρα και ο κόσμος των επιχειρήσεων αλλά και διεθνώς, ε, μιλώ για τις προκλήσεις. Λοιπόν, ε, άρα τα τελωνιακά θέματα πολλές φορές χαρακτηρίζονται από έναν έντονα τεχνικό χαρακτήρα. Ε, certains, les douanes, nous savons, le fonctionnement harmonieux euh, des douanes. Πολλές φορές δυσκολεύει την αρμονική λειτουργία αυτού του πολύ σημαντικού παρόλα αυτά πυλώνα για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει πάντοτε λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή ήταν και η βασική επιλογή που είχαμε κάνει όταν θελήσαμε να εξυγχρονίσουμε και να επεξεργαστούμε τον τελωνιακό κώδικα. Θέλαμε τα τελωνία να είναι πιο αποτελεσματικά, αποδοτικά, καλύτερες επιδόσεις για καλύτερη λειτουργία της αγοράς, προστασία των αγορών και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ο τελωνιάς κώδικας της Ένωσης που περιλαμβάνει κανόνες και υποχρεώσεις που πρέπει να εφαρμόζονται και να επιβάλλονται στους συγκεκριμένους φορείς και στις τελωνικές αρχές των κρατών μελών Ε, χαρακτηρίζεται από αποκλήσεις και διαφορές σε κάποιους τομείς εφαρμογής. Και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Όταν λοιπόν ε, δουλέψαμε πάνω στον τελωνιακό κώδικα, είδαμε τρεις βασικές κινήσεις, αν θέλετε. Θέλω να σας τις υπενθυμίσω. Όχι απλά για να επενθυμίσω την κοινή μας δουλειά, αλλά γιατί αυτοί οι τρεις κινήσεις και αυτοί οι τρεις στόχοι πιστεύω ότι θα πρέπει να μας εμπνεύσουν και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες για το έργο το οποίο θα πρέπει να ολοκληρώσουμε για αυτό το σχέδιο οδηγίας που έχει προταθεί. Πρώτη κίνηση, αν θέλετε, λισαβονοποίηση, δηλαδή ε, συμμόρφωση προς τις διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνη. Εξυγχρονισμός, δεύτερον, εξυγχρονισμός των χρησιμοποιούμενων τεχνικών και διαδικασιών κτλ. Και, και τρίτον, απλούστευση. λισαβονοποίηση, απλούστευση, εξεχρονισμός. Αυτές οι τρεις κινήσεις θα επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να μας εμπνέουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις ε, των κανόνων και των υποχρεώσεων ε, που περιλαμβάνονται στον Τελωνιακό Κώδικα της Ένωσης και σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις που θα πρέπει να επιβληθούν. Θεωρώ σημαντικό να συμπληρώσουμε κάπως για να δώσουμε μεγαλύτερη ορμή και όθηση σε αυτό το λιγνιακό κώδικα έχοντας πάντα κατά νου τις τρεις κινήσεις, τους τρεις αυτούς στόχους που μας είχαν εμπνεύσει και κατά το παρελθόν. Η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέστησε σαφέστατες αυτές τις ε, αποκλήσεις αρκετά σημαντικές που βλέπουμε μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων, μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Μέχρι στιγμή δεν έχει υπάρξει εναρμόνιση στην εφαρμογή των κυρώσεων. Επενθυμίζω ότι ο τελωνιακό κώδικα τη Ένωση που πρέπει πάνω να δουλέψουμε, και μιλάω για τι κυρώσει εδώ, αναφέρει την ανάγκη να υπάρχει αναλογικότητα, αποτελεσματικότητα και αποτρεπτικό χαρακτήρα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των κυρώσεων. Τούτων λεχθέντων βέβαια πόρο απέχουμε στην πράξη από την εφαρμογή ακριβώς αυτών των κριτηρίων. Αυτές οι αποκλήσεις, πώς εφαρμόζονται δηλαδή οι κυρώσεις, πώς επιβάλλονται οι κυρώσεις, είναι ένα θέμα που ε, γύρει δυσκολίες και είναι πραγματικά μια ανησυχία για τη συνεκτικότητα και αποτελεσματικότητα των των ελληνικών δικασιών του Τελωνιακού Κώδικα και υπάρχει πρόβλημα να έχουμε διαφορές μεταξύ των εγκεκριμένων οικονομικών ε, φορέων. Εγώ πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες, επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να υπενθυμίσουμε την προσήλωσή μας σε αν θέλετε μία ευθυγράμμιση της τελωνικής πολιτικής προς τα άνω όμως. Έχουμε <clears throat> υπόψη μας ότι με μια πιο ισχυρή εναρμόνιση πρέπει πάντα να έχουμε και μεγαλύτερο επίπεδο προστασίας των αγορών μας των προϊόντων μας, αλλά να υπάρχει και μεγαλύτερη προβολή και διαφάνεια και αποτελεσματικότητα των τελωνιακών διαδικασιών και στο σκέλος της ε, επιβολής και εφαρμογής κυρώσεων. Επομένως, κατά την άποψη μου πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, ε, θέλοντας να είμαστε συνεπείς σε σχέση με το έργο που έχουμε ήδη επιτελέσει και στόχος μας είναι από τη μια κοινοβουλευτική περίοδο στην άλλη να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις εργασίες. Και επαναλαμβάνω, δεν θα μπει σε λεπτομέρειες το ψήφισμά μας, άρα ολοκληρώνοντας σας αναφέρω κάποια σημεία που ίσως μας δημιουργήσουν κάποια προβλήματα ή τέλο πάντων να είναι αμφιλεγόμενα και να υπάρξει συζήτηση για αυτά. Πρώτον, νομική βάση. Υπάρχει συζήτηση ε, τη νομική βάση που θα ε, επιλογεί για αυτή την πρόταση πρέπει να τη συζητήσουμε ίσως και να τη συμπληρώσουμε και θα πρέπει να εγγύψουμε και στα περιθώρια λιγμών που θα πρέπει να έχουν τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του κειμένου εάν ε, ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Επίσης θα πρέπει να μελετήσουμε για μια ακόμη φορά γίνεται και στο κείμενο βέβαια αλλά πρέπει όλα αυτά να τα μελετήσουμε ξανά και ιδίω στις σχέσεις μεταξύ ε, και των χρηματοοικονομικών συμφερόντων, της νομοθεσίας που ισχύει και που πρέπει να εφαρμόζεται και τον EBC Nidem, το διπλό αξιόπινο, αυτή την αρχή που είπατε. Όλα αυτά πρέπει να τα ε, σταθμίσουμε και να τα μελετήσουμε. Και νομίζω πρέπει να έχουμε και μια σφαιρική προσέγγιση, πρέπει να έχουμε υπόψη μας κάποιες αρχές και ε, η θέση της Επιτροπής εσωτερικής αγοράς πρέπει να γίνει ξεκάθαρη για να αφήσουμε και στους διαδόχους μας ένα ισχυρό μήνυμα. Well, thank you very much for... Σας ευχαριστώ πολύ. Θέσατε πολλά ζητήματα για το θέμα της νομικής βάσης. Ίσως χρειαστεί να έλθουμε σε επαφή με τους συναδέλφους μας από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Θα γίνει ίσως μέσω της γραμματείας, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Η Εύλιν Γκέπχαρτ τώρα. Yeah, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποβολή αυτού του κειμένου και νομίζω ότι πράγματι έχει νόημα να κάνει κανείς κάποιες σκέψεις εν σχέση με τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε εσείς εδώ. Και φαντάζομαι ότι οι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους κυρώσεις οι οποίες ε, προβλέπονται εδώ και τα διάφορα ε, ζητήματα που γέρονται θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα εμπόδιο στο πλαίσιο της μεγάλης εσωτερικής αγοράς γιατί υπάρχουν ε, σημαντικές διαφορές που έχουν σαν αποτέλεσμα εκείνοι οι οποίοι θέλουν να δράσουν εγκληματικά βεβαίως θα εκμεταλλευτούν αυτές τις διαφορές μεταξύ των χωρών μελών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μεριμνήσουμε ούτως ώστε να μην γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης η εσωτερική αγορά. Γι' αυτό είναι σημαντικό που έρχεται στο τραπέζι αυτή η πρόταση οδηγία. Εσείς ο ίδιος είπατε ότι σκεφτήκατε κατά πόσο ένα, μια οδηγία ή ένας κανονισμός θα έπρεπε να επιλεγεί. Και νομίζω ότι έχετε δίκιο όταν λέτε ότι επιλέξατε τελικά τη λύση μιας οδηγίας, γιατί πράγματι οι διαφορές μεταξύ των χωρών μελών είναι τόσο μεγάλες που δεν είναι δυνατόν διαμιάς να τα συνοψίσει κανείς όλα και να πει ότι ισχύει ένα νέο ευρωπαϊκό δίκαιο χωρίς να ισχύουν αυτό το οποίο πράττουν οι χώρες μέλη. Αυτό θα ήταν ε, μια μεγάλη πρόκληση εναντί των χωρών ε, μελών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε εδώ την ευελιξία που παρέχει μια οδηγία και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε εδώ. Τώρα, σε σχέση με αυτό το οποίο προωθούμε συνήθως στο κοινοτικό δίκαιο, δηλαδή το να λέμε ότι προβαίνουμε σε μια σταδιακή εναρμόνιση χωρίς να επιβαρύνουμε υπερβολικά τις χώρες μέλη. Θεωρώ ότι σε αυτό το πεδίο του ποινικού δικαίου αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Γιατί εδώ πράγματι υπάρχουν ε, αντίθετα μεταξύ τους ε, ε, ένομα ενδιακά συστήματα. Και νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Λεγκρυπ μετά όσα είπε. Πράγματι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρόκειται να συζητήσουμε. Και παράλληλα με τα θέματα που ανέφερε ήδη η κυρία Λεγκρίπ και τα οποία δεν θέλω να επαναλάβω γιατί συμφωνώ απολύτως μαζί σας κυρία Λεγκρίπ, υπάρχει ένα θέμα που συνδέεται με το άρθρο 15 και όπου θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε ότι πράγματι μπορούν τα πράγματα να λειτουργήσουν έτσι όπως το προτείνεται όσον αφορά την δικαιοδοσία ή δεν θα είχε μάλλον νόημα στον τομέα αυτό να προχωρήσουμε έτσι όπως προχωρήσαμε και με τα άλλα νομικά ζητήματα. Δηλαδή να οργανώσουμε έτσι το ζήτημα της δικαιοδοσίας ούτως ώστε να μην λέμε ότι η χρονική στιγμή στην οποία ε, ξεκίνησε μια διαδικασία σε μια χώρα μέλος είναι και η χρονική στιγμή που ξεκινούμε εμείς αλλά να βασιστούμε μάλλον στην ίδια την παράνομη πράξη, την αξιόπινη πράξη όχι δηλαδή όπως προτείνετε εσείς να είναι καθοριστική η θαγένεια του προσώπου ή η χώρα στην οποία διαπράχθηκε το αδίκημα, αλλά το κράτος το οποίο διακινήθηκε το εμπόρευμα. Ε, ίσως θα μπορούσατε να μου δώσετε κάποιες εξηγήσεις σε αυτό το άρθρο 15, γιατί δεν κατάλαβα πολύ καλά πώς θα πρέπει να λειτουργήσει αυτό στην πράξη. Αλλά αυτή είναι μόνο μια λεπτομέρεια. Δεν θα πρέπει να απαντηθεί αμέσως γιατί κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας δεν θα έχουμε καν το χρόνο να σχολιάσουμε έτσι την σχετική νομοθεσία, όπω θα ήταν αναγκαίο. Η κυρία Λεγκρίπ και εγώ στις προπαρασκευαστικές εργασίες συζητήσαμε το με ποιο τρόπο θέλουμε στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας να προχωρήσουμε. Και εδώ τέθηκαν δύο εναλλακτικέ λύσεις. Δηλαδή, να επεξεργαστούμε να, να προετοιμάσουμε μάλλον ένα έγγραφο εργασίας ή ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και συμφωνήσαμε ότι θέλουμε να προτιμήσουμε το ψήφιμα, γιατί ένα έγγραφο εργασίας είναι, δεν είναι δεσμευτικό. Είναι μία δήλωση δύο εισηγητριών, η ενα ψηφισμα του ευρωπαικου κοινοβουλιου και συμφωνησαμε οτι θελουμε να προτιμησουμε το ψήφισμα γιατι ενα εγγραφο εργασιας ειναι δεν επικυρώνεται από κανέναν απολύτως, ενώ σε ένα ψήφισμα το οποίο βεβαίω είναι πολύ πιο βραχυπρόθεσμο. Ε, μπορούμε να επεξεργαστούμε μια πρόταση την οποία οι συνάδελφοι πράγματι θα μπορέσουν να σχολιάσουν. Και αν μπορούμε θα μπορέσει ενδεχομένω να ψηφιστεί και στην Ολομέλεια του Απριλίου. Και πραγματικά αυτή θα ήταν μια πιο δυνατή απάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω συνεδρίες των συντονιστών σήμερα να ακολουθήσουμε ακριβώς αυτήν την οδό του ψηφίσματος και αυτό θα σήμαινε ότι όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να κινηθούμε ως εξή. Το ψήφισμα θα το προετοιμάσουμε μόνο στα αγγλικά. Θα παρακαλέσουμε λοιπόν τους συναδέλφους να το αποδεχθούν στα αγγλικά. Δεν είναι τόσο το, σύντομο χρονικό διάστημα να γίνουν και μεταφράσεις γιατί ε, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο της Ολομέλειας του Απριλίου. Δηλαδή να απευθύνουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος προς τους σκιώδες και τις πολιτικές ομάδες 17 Φεβρουαρίου με την παράκληση να διατυπωθούν τα σχόλια μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου, ώστε στην Επιτροπή να μπορέσουμε στις 3 Μαρτίου να ψηφίσουμε και να συμπεριλάβουμε το ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίας Ολομελίας του Απριλίου. Αυτή είναι η πρότασή μας. Νομίζω ότι είναι εφικτό. Ήδη ξεκινήσαμε τις εργασίες μας. Θα δουλέψουμε γρήγορα. Νομίζω ότι έχει πραγματικά νόημα να τα κάνουμε έτσι τα πράγματα και περιμένω με ανυπομονησία τα δικά σας σχόλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Κέπχαρτ ε, που ορίσατε τη διαδικασία ε, και τα σχόλια. Συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι ένα ψήφισμα θα ήταν πιο ικανοποιητικό και θα υπάρχει το πλεονέκτημα να φέρουμε την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο, να παρουσιάσει σε μια πρώιμη φάση τα, τις δικές της προτάσεις και νομίζω αλλιώς θα ενισχύσουμε τη θέση της ε, Επιτροπής γιατί νομίζω ότι θα, είναι σαφές ότι θα υπάρξουν αντιπαραθέσεις μεταξύ χωρών μελών γιατί γίνονται θέματα όταν προσπαθούμε να εναρμονίσουμε τις κυρώσεις και θα είναι ευαίσθητο θέμα και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και χρειαζόμαστε μια πολιτική υποστήριξη. Ωραία λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα μέχρι ε, την ψηφοφορία. Η κυρία Ρούντερ και... Ρούλε, συγγνώμη, κυρία Ρούλε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τις προτάσεις και πιστεύω ότι το ψήφισμα πραγματικά ε, θα πρέπει να προτιμηθεί. Παρόλο που υπάρχει το εξή πρόβλημα. Από τη μία θεωρώ ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι αναγκαία και δικαιολογημένη γιατί κατέστησε σαφές ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών μελών και βεβαίω αυτό οδηγεί σε στρεβλώσει του ανταγωνισμού, σε οικονομικέ συνέπειε κλπ. Από την άλλη πλευρά, πάντοτε όταν δοκιμάζει κανεί κάτι καινούργιο, αντιστάσει είναι ιδιαίτερω μεγάλε. Και για παράδειγμα, εδώ έλαβα ένα έγγραφο των οικονομικών κύκλων της Γερμανίας που ανθίστανται κατά τις προτάσεις αυτής και θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες ε, επιστολές και δηλώσεις. Ε, λυπούμε λοιπόν που αυτή η πρόταση διατυπώθηκε πολύ αργά, θα ήταν πολύ καλύτερο εμείς ως Κοινοβούλιο να είχαμε ασχοληθεί ήδη με τα περιεχόμενα νωρίτερα. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα γιατί θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο εκκράσεων. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να χαιρετήσουμε συνολικά την προσπάθεια να γίνει επιτέλους ένα βήμα. Ε, παραπάνω από αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί αν θέλουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες θα πρέπει να κάνουμε διαβολεύσεις με εκείνους θα πρέπει συνέχεια να το εφαρμόσουν και δεν φτάνει απλούστατα ο χρόνος για να γίνει κάτι τέτοιο. I think Ο στόχος μας ήταν κυρίως για να ξέρετε τι επίκειται και όσοι συνάδελφοι έχουν ε, γνώση να μας συμβάλλουν ε, με την εμπειρία τους. Ε, εντάξει, ίσως η επόμενη όμως Βουλή μετά τις εκλογές θα αναλάβει. Κύριο Σμιτ, θέλει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε, άργησα λίγο. Αλλά ήμουν σε έναν τριμερή διάλογο που είναι σε εξέλιξη. Πάντως άκουσα μέρος τη συζήτηση και διάβασα και τις σημειώσεις ε, του βοηθού μου. Φυσικά και είναι σημαντικό το θέμα, χρειαζόμαστε κοινού κανόνες και είναι πολύ καλό. Το ότι τελικά πλέον βαδίζουμε στη σωστή κατεύθυνση Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή είναι μία προσέγγιση για τη Μολυντική Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, και ένα παλιό μου φίλο βλέπω εκεί, που ασχολείται με τα τελωνιακά. Γιατί δεν χρησιμοποιείτε για τις κυρώσεις ένα άλλο άρθρο, είναι η ερώτησή μου. Γιατί για τις κυρώσεις πρόκειται εδώ. Εσείς χρησιμοποιείτε το 33. Το 83 δεν θα ήταν καλύτερο. Δεν ξέρω αν ε, το είπε και ο πρόεδρος, ε, τέλος πάντων το υπονόησε. Είναι σημαντικό το θέμα. Η νομική βάση Αν θέλουμε πραγματικά να συμβούν ε, πράγματα, να έχουμε αποτελέσματα επιτόπου, η νομική βάση είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν η νομική μας υπηρεσία έχει να πει κάτι γι' αυτό. Εγώ πάντως πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη νομική βάση. Διαφορετικά θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο τι μπορούμε να κάνουμε. Άκουσα πάντως ε, κάποια πράγματα, διάβασα και τις σημειώσεις, άκουσα τις κυρίες Λεγκρίπ και Γκέπχαρτ και πιστεύω με όλα αυτά ότι μπορούμε να καταλήξουμε εδώ σε συμφωνία και βέβαια τώρα να ξεκινήσουμε και να ψηφίζουμε, Πρόεδρε. Πρόεδρος, να σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σμιτ. Θέλω να σας ξεκαθαρίσω το εξής. Σε καμία περίπτωση δεν πρότεινα κάποια άλλη νομική βάση, διότι δεν γνωρίζω τόσο καλά τις συνθήκες. Απλά είπα ότι υπάρχει η διαδικασία διαβούλευσης με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Δεν ξέρω αν θα έχουμε το χρόνο παρόλα αυτά. Αλλά καλό θα ήταν να στήσουμε τη γνώμη τους. Άλλοι συνάδελφοι, α, ο κύριος Κορέα, ναι, συγγνώμη, σας ξέχασα. Σας ευχαριστώ. Σύντομα, Πρόεδρε, έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Νομίζω πως είναι σημαντικό να μην προχωρήσουμε σε μεγάλες επιπλοκές όσον αφορά την ε, ε, μεταβλητή, τη μεταβλητότητα μάλλον των νομοθεσιών που ποινικοποιούν ή όχι τις παραβατικές ε, ενέργειες. Έπειτα, οι χρηματικές κυρώσεις μπορούν να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Δεύτερον, ε, μετά, εάν δεν... Ε, ναι, στο, στο μέσο της, του ψηφίσματος. Και έπειτα, έχω μια αμφιβολία, τουλάχιστον στα πορτογαλικά. Ε, γιατί το τρίτο και τέταρτο άρθρο υπάρχει η φράση πα, τελωνιακή παράβαση ή παράπτωμα και στο πέμπτο άρθρο που λέει εκ λέει παράβαση της τελωνιακής νομοθεσίας. Είναι διαφορετική έκφραση. Γιατί λέει η παρα... τελωνιακή παράβαση, ενώ στο άλλο λέει παράβαση της τελωνιακής νομοθεσίας. Είναι ηθελημένο, υπάρχει διαφορά ή είναι απλά μια έλλειψη εναρμόνιση της ορολογίας. Μάλιστα. Έχει κανείς άλλος άλλες παρατηρήσεις. Παρακαλώ να μετακινηθεί ο κάμεραμαν. Κοιτάξτε, δε, μας εμποδίζετε εκεί που στέκεστε στη μέση του κύκλου. Παρακαλώ μετακινηθείτε. Μιλώ προς τον κάμεραμαν. Yeah. Yeah, well, yes, yeah. Uh, uh, we are still discussing Συζητάμε ακόμα το θέμα. Γι' αυτό σας παρακαλώ αν θέλετε να κάνετε δικές σας συζητήσεις πηγαδάκια, ξέρω ότι πάντοτε υπάρχει μια, μια έτσι, ε, ένταση στη διάρκεια της ψηφοφορίας. Να πω ότι υπάρχουν και άλλα σημεία που αναφέρθησαν στη διάρκεια της συζήτησης. Ο κύριος Ζελίνσκη, και η κυρία όλοι θέλει να απαντήσετε, θέλετε να απαντήσετε, να σχολιάσετε αυτές τις πτυχές της παρουσίασής σας πριν κλείσουμε το θέμα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ ε, τα ε, υπόλοιπους ευρωβουλευτές της Επιτροπής. Πολύ σύντομα, οπότε κατάλαβα έχω 30 δευτερόλεπτα. Οπότε, καταρχήν, φιλοδοξία της Κομισιόν. Είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι τελικά βλέπετε, γιατί τώρα έχουμε μια προσέγγιση των ποινών. Εμείς μιλούσαμε για εναρμόνιση, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αυτά έχουμε λοιπόν ε, και θα εργαστούμε όσο γίνεται για την ε, μεγαλύτερη φιλοδοξία. Άρθρο 33 και 83. Εδώ βρισκόμαστε στο διοικητικό τομέα. Δεν θέλαμε να πούμε σε ποινικό, να φτάσουμε άλλο σε ποινικό επίπεδο, γιατί τελικά πιστεύουμε πως θα ήταν υπερβολικό για τα τελωνία. Είμαι ευχαριστημένος δε με τα σχόλιά σας. Ναι, έχουμε αργήσει, αλλά τουλάχιστον για αυτή τη θητεία, αλλά κάναμε όσο γινόταν πιο γρήγορα. Θα μπορούσα να σχολιάσω πολύ περισσότερο, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Okay. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλέ. Μάλιστα, εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Άννα Μπολή, θέλετε να πείτε κάτι. Thank you, Very briefly, 15, uh, there was a... Για το άρθρο 15 ε, τέθη ένα ερώτημα. Έχουμε ανακτήσει διάφορες περιπτώσεις που έχει κανείς τα αγαθά, ενώ υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου τα αγαθά δεν ε, μπλέκονται. Και εδώ προτείνουμε εναλλακτικά κριτήρια δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα της παράβασης, ώστε να εντοπίσουμε ποιο κράτος μέλος θα είναι αρμόδιο. Αλλά αυτό βεβαίως σημαίνει συνεργασία ανάμεσα στις αρχές των κρατών μελών. Τελευταία παρατήρηση του κυρίου Σμιτ. Συγγνώμη, από τον Πορτογάλο Ευρωβουλευτή ήταν η διαφορά ανάμεσα στην ορολογία. Στο αγγλικό κείμενο δεν έχουμε διαφορά, μάλλον είναι θέμα μετάφρασης, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχαμε πρόθεση να σημάνουμε κάτι διαφορετικό ε, και να συμπληρώσω τα όσα είπε ο κύριος Ζελίνσκι. Δεν θεωρήσαμε πως το άρθρο 83 ήταν η κατάλληλη νομική βάση, διότι η Κομισιόν δεν προτείνει ποινικέ κυρώσεις. Το συζητήσαμε αυτό με την νομική μας υπηρεσία και από ό,τι φαίνεται δεν χρειάζεται αλλά ίσως να χρειαστεί να συμπληρώσουμε την νομική μας βάση με κάποιο άλλο άρθρο, ίσως το ίδιο όπως με αυτό ε, του τελωνιακού κώδικα. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ ε, που ήρθατε και επίσης τις δύο συνεισηγήτριες που ξεκίνησαν τη διαδικασία για να ανακεφαλαιώσουμε τα όσα μας παρουσίασε η κυρία Γκέπχαρντ, ότι δηλαδή οι συνεισηγητές θα στείλουν στις πολιτικές ομάδες και στους κοιόδες εισηγητές ένα σχέδιο στα αγγλικά στις 17 Φεβρουαρίου και έχουμε υποβολή ε, τροπολογιών στις 25 Φεβρουαρίου. Μετά οι εισηγήτριες θα χρειαστεί να συναντηθούν γιατί θα χρειαστεί να ψηφίσουμε λοιπόν 3 Μαρτίου για να έχουμε και μια θέση στην Ολομέλεια. Η διαφορετικά δεν έχει νόημα να τα κάνουμε όλα αυτά, εκτός και αν έχουμε μια σωστή συζήτηση στην Ολομέλεια που θα προσπαθήσουμε, θα στοχεύσουμε την πρώτη Ολομέλεια του Απριλίου στις Βρυξέλλες. Αυτά λοιπόν. Τώρα θα προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Παρακαλώ λοιπόν να καθίσετε για να ψηφίσουμε. Να καλέσω εδώ τη γραμματεία να έρθετε να κάτσετε εδώ πίσω μου για να ελευθερωθούν και κάποιες θεσούλες εκεί. Δεν είναι η κανονική μας αίθουσα που κάνουμε τις ψηφοφορίες. Ε, τουλάχιστον οι πλειοψηφίες είναι εδώ μπροστά μου με την ότι σηκώνετε τα χέρια σας. Κάποιες θέσεις λοιπόν ε, καθαρίζουν εδώ για όσους στέκονταν πίσω-πίσω. Σας ευχαριστώ για το μεγάλο σας ενδιαφέρον ε, στην... για τις εργασίες μας. Uh, then we can get on with the voting. So, um, Για να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία λοιπόν και θα ψηφίσουμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι... Το αποτέλεσμα των άτυπων διαπραγματεύσεων, ε, τριμερών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για τις δημόσιες συμβάσεις, όπου είχαμε εισηγείται την κυρία Κόλεν Λάγκε. Σας παρακαλώ να μας παρουσιάσετε το αποτέλεσμα όλων αυτών και μετά να ψηφίσουμε μόνο μία ψηφοφορία ηλεκτρονικά για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Η κυρία Λάγκεν. Ναι, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πετύχαμε καλούς συμβιβασμούς. Το πιο σημαντικό σημείο ή μάλλον τα πιο σημαντικά σημεία ήταν τα εξής. Συμφωνήσαμε οι εκχωρήσεις να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής και συγκεκριμενοποιήσαμε τις γενικές απαιτήσει όσον αφορά την ενδετερότητα της τεχνολογίας, την προστασία των δεδομένων κλπ. Έχουμε επίσης συμπεριλάβει τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς σε ένα νέο άρθρο και δώσαμε χρόνο στην Επιτροπή ε, μάλλον περιορίσαμε το χρονικό διάστημα ε, σε 36 μήνες και εδώ εμπίπτει και ε, η δυνατότητα δοκιμών ούτως ώστε το κόστος να είναι το ενδεδειγμένο και να είναι ε, φιλικό προς το χρήση, χρήστη. Έχουμε 18 μήνες για την ε, διανομή και ε, νομίζω ότι συνολικά πετύχαμε ένα καλό συμβιβασμό και μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι που με τον τρόπο αυτό το σύνολο του πακέτου μπορεί να εφαρμοστεί ήδη στο πλαίσιο αυτής της θητείας και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία αν δούμε το σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και σένα και όλους τους σκιώδεις. Νομίζω ότι πετύχαμε με ένα εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα αν δούμε το χρονοδιάγραμμα. Ωραία λοιπόν, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τι κάνουμε, βλέπουμε τα αποτελέσματα και πάνω ή πρέπει εγώ να τα διαβάσω. Θα δείτε μπροστά σας τα αποτελέσματα, αλλά καλύτερα να τα διαβάζω κιόλα. The vote is open electronically. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Έχουμε 37 κάρτες, 34 όμως μπορούν να ψηφίσουν. Yeah. Sorry, we're just rearranging ourselves here. All uh, right, there are 37 cards in, but only... 37 κάρτες λοιπόν, 38. Θέλει κανείς άλλος να ψηφίσει. Όχι, έχουμε 38 λοιπόν. Πέρα τη ψηφοφορία και εγκρίνεται με 37 ψήφους υπέρ και μία κατά. Σας ευχαριστώ και περνάμε στην Ολομέλεια. Και ποια Ολομέλεια? Μάρτιος νομίζω. Ίσως και τη δεύτερη του Απριλίου. Εξαρτάται. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κόλιν Λάγκεν. Δεύτερο σημείο που είναι ένα τυπικό σημείο και δεν βλέπω τον κύριο Ταραμπέλα εδώ, αλλά θα το αναφέρω εγώ λοιπόν, εξ του. Ως αποτέλεσμα της λεπτομερούς εργασίας προετοιμασίας κειμένου για τις δημόσιες ε, υπηρεσίες, ε, ανακαλύφθη ένα λάθος σε ένα παράρτημα στο οποίο, για το οποίο υπήρχαν παραπομπές και το έχετε ήδη δει όλοι σα οι σκιώδει ηγητέ το έχουν εξετάσει, αλλά είναι μια τεχνική διόρθωση, αλλά πρέπει τύπη να το εγκρίνουμε. Λοιπόν, εκτό αν έχετε ερωτήσει, ε, νομίζω πω όλε οι ομάδε το έχετε συζητήσει. Θα ήθελα τύπη να το ψηφίσουμε. Λοιπόν, είναι ένα διορθωτικό ε, με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου όσον αφορά την οδηγία για τι δημόσιε συμβάσει ε, και ψηφίζουμε. Uh, please vote. If you can hurry up and vote, it would be helpful. Uh, the vote is closed. Uh, Ωραία, λοιπόν, τέλος ψηφοφορίας. 37 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία για τον κύριο Μπίλαν. Συμφωνήσαμε με τον κύριο Μπίλαν να ψηφίσουμε πρώτα αυτή την έκθεση που είναι η γνωμοδότηση του κυρίου Πίλαν για την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Δική μας γνωμοδότηση λοιπόν για τα τέλη για τις πληρωμές με χρεωστική πιστοτική κάρτα. Κύριε Πίλαν θέλετε να πείτε κάτι τώρα, όχι. Οπότε προχωράμε κατευθείαν στην ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση του κυρίου Μπίλαν. Είστε όλοι έτοιμοι. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε την τροπολογία 19 επί του τίτλου Μια οριζόντια τροπολογία του κυρίου Σαλβίνη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έξι του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 30 καταπίπτει. 31 έχει αποσυρθεί. 32 μπίλαν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. μπήλαν, Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Καταπίπτει 34 σαλαφίνι, Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35. μπήλαν, ως προστίκη. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 8 δεν την ψηφίζουμε. Συμβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. Προχωράμε στην 43 του κυρίου Σαλβίνη. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 νομίζω καταπίπτει. Έχω δίκιο. Την εγκρίναμε τη 19. Όχι, την απορρίψαμε. Ωραία. Πάμε στις 45 και 46. Υπέρ. Α, νομίζω εδώ καλύτερα ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε. 45 και 47 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται 22 κατά, 15 υπέρ. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 54 με προφορική τροπολογία του εισηγητή, την οποία βλέπετε εδώ. Ποιοι είναι υπέρ. Κύριε Σφάμπα. Όχι. Είναι σημαντικό να βρεθεί λύση για τις μικροπληρωμές, αλλά αυτό που προτείνεται δεν δίνει κάποια εξήγηση, οπότε είμαστε κατά της προφορικής. Μάλιστα. Υπάρχει μια παρεξήγηση, Πρόεδρε, γιατί ο κύριος Μπόρισοφ αναφερόταν στην προφορική που θα έπρεπε να υποβάλει ο κύριος Δε Γιόγκ, αλλά από ό,τι κατάλαβα ο κύριος Δε Γιόγκ δεν έχει υποβάλει προφορική ερώτηση. Αλλά αυτή την προφορική που είναι στον κατάλογο ψηφοφορίας μπορούμε να τη δεχτούμε. Κοιτάξτε, εγώ για ποια μιλάω. Αυτή που είναι στον κατάλογο ψηφοφορία σας, αυτή την προφορική, έχει κανείς αντίρρηση για αυτήν, όχι. Ωραία λοιπόν, να ψηφίσουμε σε αυτήν και έπειτα αν υπάρχει κάτι άλλο το, το λύνουμε μετά. Ποιοι είναι υπέρ της 54 Στάιλερ, με τη δική σας τροπολογία που είναι μέσα στον κατάλογο ψηφορής υπέρ κατά, εγκρίνεται. Υπήρχε πρόταση για μια ακόμα προφορική, αλλά που τελικά το ΕΛΚ δεν την επιμένει. Οπότε δεν χρειάζεται να τη συζητήσουμε. Ωραία. Ωραία λοιπόν τότε. Περνάμε γιατί πολλές κατέπεσαν λόγω της συμβιβαστική και σύμφωνα με τη δική μου λίστα πάμε στην ε, τροπολογία 16 του εισηγητή τώρα. Αλλά και πάλι με προφορική τροπολογία που έχετε στον κατάλογο ψηφοφορίας σας, φαντάζομαι ότι δέχεστε, οπότε έχουμε την τροπολογία 16 με την προφορική υπέρ κατά εγκρίνεται. Και έπειτα έχουμε την 70 του κ. Σμίτ ως προσθήκη. Στην 16 υπέρ κατά εγκρίνεται. 72 μπίλαν υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 17 μπίλαν με προφορική τροπολογία που βλέπετε. Υπέρ. Κατά. Α, μάλλον να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά γι' αυτό. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν γιατί είναι 17 υπέρ. Ε, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν 23 ψήφοι υπέρ, 13 κατά. Τροπολογία 73, Μπορισόφ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74, 75 έχουν καταπέσει. 76, υπέρ. Ποιοι είστε υπέρ, παρακαλώ, κατά. Νομίζω πως απορρίπτεται. Αλλά εδώ το έλκα έχει χωρίσει. Έχει διχαστεί. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 76. Ναι, αυτό βλέπω. Έχει διχαστεί, εν πάση έχει χωρίσει. Ε, λοιπόν. 20 υπέρ, 18 κατά. 77 της κυρίας Βερνιό, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 78 Μπίλαν, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 79 Βερνιό, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 80 Μπορισόφ υπέρ. Ποιοι είστε παρακαλώ υπέρ. Κατά. Ε, να ελέγξουμε. Εντάξει, να ελέγξουμε την 80 ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. 16 υπέρ 22. Είχα... Δεν είχα δίκιο για αυτήν. 81. υπέρ κατά και πάλι το ίδιο νομίζω είναι, οπότε καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, να ελέγξουμε. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. δύσκολο να πω έτσι πως ε, ε, καθόμαστε λοιπόν ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται 19-19 Ευτυχώς που έλεγξα 83 Σαλβίνη υπέρ κατά απορρίπτεται 84 έχει απορριφθεί 85 υπέρ κατά απορρίπτεται 86 υπέρ κατά απορρίπτεται 87 υπέρ κατά εγκρίνεται 88 υπέρ εγκρίνεται 89 υπέρ κατά εγκρίνεται 90 υπέρ κατά πρέπει να ελέγξουμε νομίζω 90. Ένας παραπανήσιος έλκα ψήφισε. Μάλιστα. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Τώρα περνάμε στα εισιτιολογικές σκέψη. Ένα του εισηγητή. Περ. κατά εγκρίνεται 20 υπέρ κατά εγκρίνεται 21 υπέρ ψηφίζει ναι 20 υπέρ κατά εγκρίνεται 21 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 6 Αυτομάτως εγκρίθηκε με την 5, οπότε πάμε στην τροπολογία 3 που συνδέεται με τη 16. Πρέπει να την ψηφίσουμε όμως χωριστά. Υπέρ, ποιοι είναι, κατά, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 26 συνδέεται με την 80 που έχει απορριφθεί. 5 του εισηγητή, υπέρ, κατά, Κατά. Πολύ τσίμα τσίμα είναι η ψηφοφορία. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Την 4 νομίζω την είχαμε ψηφίσει. Την 4, την 4 του εισηγητή, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 27 έχει καταπέσει. 28 και 29 δεν χρειάζεται να ψηφιστούν γιατί συνδέονται αυτόματα με προηγούμενες ψηφοφορίες και περνάμε στο σχέδιο γνωμοδότησης. Τελική λοιπόν ψήφος για το σχέδιο γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Οικονομικών. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Παρακαλώ ψηφίστε. Μόνο 35 ψηφίσατε μέχρι τώρα. Εγκρίνεται λοιπόν με 37 ψήφους υπέρ και μία κατά. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν κύριε Μπίλαν και ελπίζουμε να το προωθήσετε και στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Okay. Now, we, our next um, vote is on the report of Mrs. Senalova. Um, να περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία. Είναι η έκθεση αυτή, ξέρετε, μια έκθεση που Μα έχει απασχολήσει εδώ καιρό και με την Επιτροπή Μεταφορών και με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθερών συνεργαστήκαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα συνεδριάσαμε μακρόν για να ολοκληρώσουμε, να εντάξουμε, συγγνώμη, και παρακαλώ σιωπή γιατί είναι σημαντικό, για να ενσωματώσουμε και τι απόψει απόψεις Επιτροπή Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Έλαβα όμω μια επιστολή χθε το βράδυ από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που θεωρεί ότι οποιαδήποτε απόπειρα τροποποίησης του κειμένου που πρότεινε η ΛΥΜΠΕ και σας παραθέτω θα οδηγήσει σε απόρριψη από πλευράς και θα θεωρήσουν ότι δεν είναι έγκυρη η ψηφοφορία μας. Δεν γνωρίζω σε τέτοιο βάθος τον ιστορικό κανονισμό αν λάβουμε υπόψη τι ανησυχίε του, μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω τι θέλει ε, ε, να μα συμβουλεύσει η... ο εισηγητή και σκιώδη για να έχουμε μια ξεκάθαρη θέση. Κυρία Σενάλο Βελκού, να μας πει τι, τι πιστεύει. Πρόεδρε, είπατε ακριβώς τι προσπαθήσαμε να κάνουμε. Ο στόχος μας ήταν να ενσωματώσουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ στο προτινόμενο κείμενο. Για να είναι ένα κείμενο συνεκτικό, πλήρες και να ανταποκρίνεται στους στόχους αυτού του κανονισμού. Είπατε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε μια μακρά συνεδρίαση με τους κοιότητες εισηγητές εξετάσαμε τις ε, μεμονωμένες προτάσεις της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και με βάση τα επιχείρηματά τους και τις προτάσεις τους καταλήξαμε σε ένα συμπεριβαστικό κείμενο που θα αποτελέσει και αντικείμενο της ψηφοφορίας σήμερα. Η γνωμοδότηση, μάλλον η άποψη της διάσκεψης των Προέδρων δεν μας βοηθά να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι η κατανόμη των αρμοδιοτήτων. Εγώ λοιπόν θα έλεγα να ψηφίσουμε την έκθεση όπως έχει υποβληθεί και οι πολιτικές ομάδες να αποφασίσουν μετά η καθεμία πώς θέλουν να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Αυτό υπερβαίνει τις δικές μου αρμοδιότητες ως, ως εισηγήτριας, αλλά και τις συμβαστικές προτάσεις στις οποίες εγώ κατέληξα. Εγώ λοιπόν προτείνω να ψηφίσουμε την έκθεση όπως έχει υποβληθεί. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεγιόγκ θέλει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι στην ευτυχή θέση να έχω και εγώ συμμετάσχει στην σύνταξη της γνωμοδότησης ΦΟΣ, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ δηλαδή. Και παρακαλώ πραγματικά την Επιτροπή σας, ναι, φυσικά και μπορείτε να πιέσετε, να αγκριθείτε οτιδήποτε. Όμως, εγώ πιστεύω ότι η έκβαση αυτή της ψηφοφορία δεν θα είναι αποδεκτή, τουλάχιστον για τη δική μου πολιτική ομάδα, αλλά νομίζω και για άλλες πολιτικές ομάδες, δεν θα είναι λοιπόν αποδεκτή ως διαπραγματευτική βάση. Ας είμαστε ενήλικοι εδώ στην Επιτροπή μας. Αν υπάρχουν δύο επιτροπές που έχουν κάποιο πρόβλημα, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και προσπαθούν να, βρουν μια φιλική λύση. Προτείνω λοιπόν να μην ψηφίσουμε τώρα, αλλά πρώτα οι συγητές να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση. Πρόεδρος. Ήρθε ο κύριος Βος τελευταία στιγμή και δεν τον καλωσόρισα. Ο κύριος Φως λοιπόν ήταν εισηγητής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθερίων. Ήταν εξαιρετική η σχέση και η συνεργασία που είχαμε, το τονίσω αυτό. Πείτε μας κύριε Βος την άποψή σας, τι μας προτείνετε και μετά θα προσπαθήσω να πιάσω και τον σφιγμό της Επιτροπής μας για να δούμε τι πρεσβεύουν. Κύριος Βος. Ευχαριστώ πολύ και για τη δυνατότητα που μου δώσετε να εκφραστώ εδώ εν συντομία. Όταν σε ένα ντοσιέ υπάρχει μέσα το σκουλίκι, τελικά παραμένει το πρόβλημα. Ε, με τον εισηγητή θεωρώ ότι βρήκαμε πολύ καλές δυνατότητες, αλλά στη συνέχεια υπήρξε μια συναισθηματική φόρταση, η οποία κλιμακώθηκε στο επίπεδο των σκιωδών καθώς και των Προέδρων των Επιτροπών, κάτι το οποίο πραγματικά είναι ιδιαίτερο ατυχές για αυτό το ντοσιέ. Το θέμα του πώς ερμηνεύει κανείς το Rule 50, νομίζω ότι θα πρέπει να το διευκρινίσουν οι επικεφαλείς των ε, επιτροπών. Εγώ ίδιος είμαι διατεθειμένος να συμπεριλάβω αυτές τις ε, τεχνικές ε, αλλαγές στο κύκλο των σκιωδών κάτι που μέχρι στιγμής δεν μπόρεσε να γίνει. Αλλά ε, πραγματικά θα ήμουν πολύ κατά ε, τελικά να δημιουργηθούν μέσω ψηφοφοριών κάποια τετελεσμένα ε, ή δεδομένα χωρίς να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι ακριβώς τα περιεχόμενα των επιμέρους σημείων γιατί θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε αυτή την παραλλαγή αλλά αν υπάρχουν συναισθηματικές ε, φορτίσεις και μείνει η ΛΥΜΠΕ ε, στο άρθρο 6 και την ε, σχετική αιτιολογική σκέψη, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Νομίζω θα πρέπει να υπάρξει μια διευκρίνηση ως προς τα περιεχόμενα και να δώσουμε χρόνο για αυτό το κείμενο ώστε να συμφωνήσουμε επί της διαδικασίας που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Ωραία. Νομίζω... Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε ε, και νομίζω ότι πραγματικά ίσως θα ήταν καλό να προετοιμάσετε από κοινού μαζί μας μια λογική πρόταση για την Ολομέλεια. Αλλά να δούμε τι θα κάνουν και οι άλλες ε, ομάδες. Ο κύριος Μάντες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι εμείς ως Επιτροπή ε, εδώ έχουμε τη δική μας ευθύνη, αλλά έχουμε και την Ολομέλεια και έχουμε μια κοινή ευθύνη και με τις άλλες Επιτροπές. Γι' αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να το ψηφίσουμε αυτό το σημείο εδώ ως Επιτροπή ε, Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και ε, εάν είναι δυνατόν να ξεκινήσουν οι συζητήσεις τριμερούς επίπεδου να συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Προετοιμάστε την θρολομέλεια. Να κάνουμε δηλαδή την ψηφοφορία, αλλά στη συνέχεια με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με τις άλλες ε, επιτροπές. Αλλιώς θα υπάρξει χάος στην Ολομέλεια. Η ε, κυρία Βαντεκάμπ. Ε, ναι, κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω στα αγγλικά για μία φορά, αλλά ποτέ, ο κύριος ποτέ πια ξανά. Ε, και σε αυτό το σημείο συμφωνώ με το κύριο Μάντες. Όπως είπατε, καθώς και ο κύριος Βος και ο κύριος Ντε ε, έχουμε πίσω μας μακρές διαπραγματεύσεις για αυτό το ντοσιέ. Και δεν πρόκειται μόνο για το πρόβλημα με τη Λίμπε, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο συζητάμε εδώ και δέκα χρόνια και νομίζω ότι τώρα στο τέλος αυτής της θητείας θα πρέπει να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτή τη συζήτηση και να αξιοποιήσουμε το χρόνο μεταξύ ψηφοφορίας Επιτροπής ΙΜΚΟ και Ολομέλειας ε, να πετύχουμε μια συμφωνία με τον κύριο Βός και τους Σκιώδης. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, καθώς και ο κύριος ε, Βός το ίδιο. Και οι Σκιώδης επίσης. Ο Σβάμπ επίσης το καταλαβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνάντηση των σκιωδών ε, κατέστησα σαφέ ότι η δική μου πολιτική ομάδα έχει πολλές επιφυλάξεις προ το θέμα αυτό. Ποτέ δεν είμαστε υπέρ ε, να γίνει υποχρεωτικό το e-call. Αλλά χάσαμε εδώ και αποφάσει που έχει χάσει κανεί. θα πρέπει να τι αποδεχθεί και δεν θα πρέπει μέσω κόλπων να προσπαθεί εκ των υστέρων να τι ακυρώσει. Γι' αυτό νομίζω ότι κάναμε τα πάντα για να κάνουμε καθαρέ διαπραγματεύσει και θα έπρεπε τώρα να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ε, Βεβαίω, πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, θα συζητήσουμε με τη ΛΥΜΠΕ και τι άλλε επιτροπέ. Αλλά αυτό δεν είναι ζήτημα, αλλά και η ΛΥΜΠΕ θα πρέπει επίση να σεβαστεί τι διαδικασίε. Και είχαν ε, προηγουμένω αρκετέ ε, ευκαιρίε και θα έχουν και μια άλλη ευκαιρία πριν από την Ολομέλεια. Να νομίζω ότι μέχρι εδώ όλα αυτά αρκούν. Um, ε, λοιπόν, νομίζω, ότι, καταρχήν μάλλον έχω την εντύπωση ότι βεβαίως υπάρχει διαχωρισμό. Ο κύριος Βαντεκάπ και η κυρία Αναλόβα είναι απολύτως ξεκάθαρες ότι θέλουν να προχωρήσουν στην ψηφοφορία των προτάσεων. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές και με τον κύριο Βος ότι στη συνέχεια θα είμαστε ανοιχτοί δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια. Δεν βλέπω αυτό να είναι πρόβλημα. Και νομίζω ότι είναι σαφές από τον κανονισμό ότι όταν υπάρχουν κάποιες ε, επιφυλάξεις και το άρθρο 30 αφορά ακριβώς τομείς ε, όταν ένα θέμα άπτεται των αρμοδιοτήτων δύο ε, επιτροπών. Δεν είναι αυτή η περίπτωση εδώ, κύριε ε, πρόκειται για το, την περίοδο έγκρισης αυτών των οχημάτων. Ε, νομίζω ότι είναι σαφές ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε στην επίτευξη ενός αποτελέσματος μέσω συνδιαλλαγής. Και νομίζω ότι η θέση των εισηγητών με εξαίρεση τον κ. Τεγιόγκ είναι να ψηφίσουμε το κείμενο του συμβασμού προτάθηκε από τον εισηγητή το οποίο λαμβάνει υπόψη του πλήρως την Επιτροπή της ΛΥΜΠΕ όσον αφορά την ουσία, όχι ίσως ως προς την ακριβή διατύπωση. Ε, αν θέλετε λοιπόν θα πρέπει να πάμε στην ε, συνδιαλλαγή μετά ούτω ώστε να έχουμε την υποστήριξη της ΛΥΜΠΕ στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι αυτή είναι μια λογική προσέγγιση και χαίρομαι θα μπει στα πρακτικά εκ μέρου τη Επιτροπής. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια λογική τοποθέτηση. Στο βαθμό όμως... Ε, ε, ε δεν ξέρω, αυτή την θέση θα ακολουθήσουμε. Δεν ξέρω, θέλετε να επανέλθετε σε αυτό το θέμα. Παρακαλώ να με συγχωρέσετε και πάλι. Ωστόσο, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ την κατάσταση του Rule 50, του κανονισμού 50, αυτό το οποίο ψήφισε η ΛΥΜΠΕ ε, έστω και αν δεν είναι βολικό ως προς τα επιμέρους σημεία, ε, ε, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό. Το άρθρο 6 και τη λογική σκέψη 13 θα πρέπει να παραμείνουν έτσι όπως ε, τις ψηφίσαμε. Γι' αυτό θεωρώ ότι όσο αφορά τη διαδικασία θα ήταν καλύτερο καταρχήν να φτάσουμε σε μια συμφωνία και μετά να περάσουμε στην ψηφοφορία. Αλλά αν εσείς πάρετε μια άλλη απόφαση τότε όσον αφορά το Rule 50 ε, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το δικό μας κείμενο, αλλά θα πρέπει να το πάρουμε ως έχει. Έτσι τουλάχιστον κατανοώ εγώ τον κανονισμό. Well, I mean, I think... Ακούστε. Είναι θέμα δύσκολο, σίγουρα. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε αντιπαράθεση με άλλες επιτροπές. Το θέμα παραμένει όμως ότι εμεί λάβαμε πλήρω υπόψη τις δικέ σα τροπολογίε. Όλες σα τις τροπολογίε τι ενσωματώσαμε στο κείμενό μας. Πλευράς λοιπόν ποιότητα τη νομοθεσία είναι καλή έκβαση. Εμείς είμαστε ουσιαστικά ε, η αρμόδια. Δεν υπάρχει απόλυτη ισορροπία μεταξύ των αρμοδιοτήτων των επιτροπών. Νομίζω ότι αυτό το άρθρο ε, Μπορεί να μην ήταν ε, το κατάλληλο, αυτό εφαρμόζει η διάσκεψη των πρόεδρων για αυτή την έκθεση. Εμείς ε, δαπανίσαμε πολύ χρόνο για να εξετάσουμε όλες, μας τις, όλες σας τις τροπολογίες και με την Επιτροπή Μεταφορών, ε, την άμεση του 49, εργαστήκαμε πολύ καλά. Έχοντας όλα αυτά υπόψη, ε, καταλαβαίνω την άποψη και τη θέση της εισηγήτριας. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Η εισηγήτρια η Σκιώδης ε, από το ΕΛΚΑ και, και ο Σκιώδης από τους Πρασίνους. Ε, αυτό θέλουν να γίνει. Ε, Δυστυχώ δεν έχω άλλη επιλογή παρά να έτσι να προχωρήσω κύριε Βόσο, κύριο ε, Μάντερ. Μία λύση κύριε Πρόεδρε, να ψηφίσουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας, αυτό το κείμενο που έχουμε μπροστά μας και βέβαια πάντοτε είναι δυνατό ε, για το άρθρο 6 και για 13 που εγκρίθηκαν στη ΛΥΜΠ να επανακαταθέσουν τροπολογίες όσοι συνάδελφοι θέλουν στην Ολομέλεια. Πρόεδρος, ναι πράγματι, αυτό πάντοτε είναι μια δυνατότητα, έτσι ισχύει και έτσι με αυτή τη βάση μπορούμε να προχωρήσουμε. Να έχουμε όλοι όμως υπόψη μας τις συνέπειες. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών τότε μπορεί να θελήσει να αμφισβητήσει την ψηφοφορία μας, να τη θεωρήσει άκυρη και να ζητήσει να ξαναψηφίσουμε από την αρχή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αναπόφευκτα θα ε, αργήσουμε πάρα πολύ και δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε πριν τη λήξη της θητείας αυτού του Κοινοβουλίου. Να έχουμε υπόψη μας ποιες είναι οι συνέπειες λοιπόν. Από πρακτικής πλευράς και φαντάζομαι θα συμφωνήσει και ο κύριος Βός, εμείς αυτό που θελήσαμε ήταν να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους καταναλωτές και για την ασφάλεια το, την οδική. Ε, αυτός ήταν ο στόχος, ο βασικός. Ειλικρινά σας το λέω δεν θα περιποιήσουμε τιμή στην ε, εικόνα του Κοινοβουλίου αν εργαστούμε αυτόν τον τρόπο και αν κάνουμε αυτά τα πισωγυρίσματα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούσαμε για να σωματώσουμε τις προτάσεις της Επιτροπής Λίμπε στην δική μας έκθεση. Εγώ δεν βρίσκομαι εδώ σταματοφύλακα των κανόνων, αλλά ερμηνεύοντας τους κανόνες θεωρώ ότι αυτό που κάνουμε είναι απολύτως αποδεκτό. Όμως, Όπως είπα, είμαστε αδιαμφισβήτητα η καθήλα αρμόδια επιτροπή, γιατί είναι θέμα εσωτερικής ενίας αγοράς, είναι δική μας αρμοδιότητα, δεν υπάρχει γι' αυτό κάποια αμφισβήτηση. Άρα οι διαδικασίες του άρθρου 50 και θα έλεγα σε αντίθεση με το τηλεπικοινωνιακό πακέτο που εκεί με την Επιτροπή Βιομηχανίας είχαμε, είμαστε σε ανισότιμη θέση. Εδώ δεν ισχύει αυτό. τα θέματα δεδομένων, προστασίας δεδομένων, επιτροπή ΛΥΜΠΕ, είναι εμένα συνδεδεμένα, πρέπει να ενταχθούν στο συνολικό πακέτο για να είναι λογικό και να λειτουργήσει σωστά. Και συμφωνούν όλοι. Και νομίζω όμω ότι το έχουμε πετύχει και μπορούμε από πλευρά ποιότητα νομοθεσία να θεωρήσουμε ότι είναι αποδεκτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, άρα προχωράμε, ψηφίζουμε. Προπολογές 34 και 35. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 1 του της εισηγήτριας, ψήφι Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 64, De Jong, ψήφι Κατά. Απορρίπτεται. Ήταν το ιδέσμι 1. Πάμε στη συμβιβαστική τροπολογία 26, κατά τμήματα, όπως ζήτησε η Άλντε. Πρώτο τμήμα, Χωρί τις λέξει and agricultural tractors υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα για την προσθήκη αυτών των ε, λέξεων και γεωργική ελκυστήρες υπέρ κατά εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Περνάμε λοιπόν τώρα στη συμβιβαστική 12, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 της ηγήτριας, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Οι επόμενε τροπολογίε καταπίπτουν και περνάμε στη συμβαστική 13. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνει. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 15 τη ηγήτρια. και τη 10 η Ήτρε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Λίμπε 9. Α, θα το δούμε μετά. Όταν φτάσουμε στη Λίμπε 10. Συμβιβαστική 16. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τραν 18 ψηφιπέ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16 και Ήτρε 12 ψηφιπέ, Κατά. Εγκρίνονται. Τροπολογία 17 της και Ήτρε 13 ψήφι Κατά. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Τραν 19, 18, 14 και τα λοιπά και 19 της υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Ήτρε 15. Καταπίπτει. Τροπολογία 72 είχε αποσυρθεί, είχε απορριφθεί μάλλον, άρα έχουμε την τροπολογία 20 και την Ήτρε 16 υπέρ. Κατά εγκρίνονται. Τροπολογίες 75, 73, 74 καλύπτονται από συμβιβαστικές Συμβιβαστική 14 ψήφι υπέρ, κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 ψήφι υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τραν 22. Καταπίπτει. Ναι. Άρα πάμε στην συμβαστική 23. Υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. και 79. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ε, απορρίπτεται. 80 καταπίπτει νομίζω ή όχι. Μάλιστα, καταπίπτει. Συμβιβαστική 17. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Τι έγινε με αυτήν. Κατέπεσε ή όχι. Μισό λεπτό να ελέγξουμε τι γίνεται. Όχι, θα την ψηφίσουμε την τροπολογία 25 της ψήφι ψήφιπε. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Ψήφι υπέρ. Με την προφορική τροπολογία του κυρίου Μάντερ, συγγνώμη. Κύριε Μάντερ, είναι, είναι στον κατάλογο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριος Μάντερς. Το ΕΛΚ είχε ζητήσει διαγραφή της λέξης vehicle, οχημάτων. οχημάτων. Αν όμως ε, ε, το καταργήσουμε, θα έχουμε πρόβλημα με τα συνεργεία. Εγώ νομίζω καλό είναι να επαναλαμβάνουμε για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Πρέπει αυτή τη λέξη μα για τους μικρούς ε, μηχανικούς, τα μικρά συνεργεία, να το αφήσουμε αυτό το, αυτή τη λέξη Το δέχεστε κυρία Σενάλοβα, λέει ο πρόεδρος, όχι. Δεν υπάρχει συμφωνία για την προφορική τροπολογία. Η κυρία Σενάλοβα, η συγγήτρια, είναι αντίθετη. Φαντάζομαι όλη η ομάδα των σοσιαλιστών, γιατί χρειάζονται και άλλοι δύο, είναι αντίθετη. Άρα θα ψηφίσουμε χωρί την προφορική τροπολογία. Συμβαστική δεκοτό χωρί την προφορική υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα, πού πάμε. Στη συμβαστική 20 πάμε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε πάλι παρακαλώ. Υπέρ τη 20. Κατά. Μάλιστα, εγκρίνεται. Ξεκάθαρο ήταν. Την 28 πρέπει να την ψηφίσουμε τη ηγητρίας. Ναι. Την ψηφίζουμε. 28 της ηγητρίας, γιατί είναι συμβατή με όλα τα άλλα. Από ό,τι βλέπω, ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21, ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 102. De Jong. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Λίμπε 10 καταπίπτει. 102. Μάλιστα. Την 102. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Α, θέλετε να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Μάλιστα. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Αν και νόμιζα ότι είχε αποσυρθεί. Απορριφθεί, συγγνώμη. Εσεί θέλετε να ξέρετε τη διαφορά των ψήφων από ό,τι βλέπω. Ορίστε, απορρίπτεται. 6 ψήφι 5, 31 κατά. Λοιπόν, προχωρούμε στην τροπολογία 32 της εισηγήτριας. 32 της εισηγήτριας. Ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Πηγαίνουμε τώρα στην 105, ναι, γιατί δεν εγκρίθηκε 102. Τροπολογία 105, ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τώρα πάμε στη συμβιβαστική 24, ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική... Α, όχι. Λίμπε. Λίμπε 12. Λίμπε 12 πρέπει να την ψηφίσουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Και τώρα συμβαστική 23α ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 25 ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τραν 33 ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 113 ψήφι υπέρ κατά εγκρίνεται 114 δέσμη, δέσμη 2, ε, ψήφι υπέρ, κατά εγκρίνεται. Άρα μετά, λείπε 14 προστίκη, υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 115 έχει εγκριθεί στη δέσμη αυτή 2, άρα πάμε στην τραν 36, υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 116 και λίμπε 16 υπέρ. Κατά εγκρίνονται. Τραν 37 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 117 λίμπε 17 ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνονται. Και μετά κάποιες ε, που ακολουθούν ε, καταπίπτουν. Και περνάμε στη συμβιβαστική 27 ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Περνάμε στα στις σκέψη, τροπολογία 2 της συγκήτριας. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ήτρε 1. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ήτρε 2. Υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβα... Μάλλον τροπολογία 45. Καταπίπτει, ναι, άρα συμβαστική 4, είπε, κατά. Εγκρίνεται. Όχι, ήταν μια τμηματική ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος της ε, Άλντε. Πάμε στο πρώτο τμήμα, χωρίς του τους ελκυστήρε. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και τώρα να προσθέσουμε του ελκυστήρε. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 4 της γήτρες υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Βλέπω ότι εδώ έχουμε την προφορική τροπολογία. Φαντάζομαι ότι δεν τη δέχεστε, ε, κυρία Σενιάλοβα. Μάλιστα. Άρα, συμβιβαστική 8 χωρίς την προφορική υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 της ηγήτριας και άλλες δύο. Υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 10 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Λίμπε 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τραν 11, καταπίπτει. Συμβιβαστική 10β, 10β, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10α, 10α, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 11, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης. 38 έχουν βάλει τις ε, κάρτες. Πέρας ψηφοφορίας. Ψήφισαν 37 συνάδελφοι. Αποτέλεσμα 34 ψήφοι υπέρ. 2 κατά μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση της κυρίας Σενιαλόβα με μεγάλη πλειοψηφία. Σας ευχαριστούμε για τη δουλειά σας κύριε Σενιαλόβα. Λοιπόν, τώρα, πριν ε, φύγετε κύριε κυρία Αναλόβα, θέλετε να κάνετε μία πρόταση για μία εντελή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο στη φάση αυτή. Η αρχική μου πρόταση ήταν ναι. αλλά θα ήθελα να ακούσω τι θα πούν και οι πολιτικές ομάδες ε, κάτω από το πρίσμα των όσων ακούσαμε από τον κύριο Φως. Κατά πόσο μας σε θέση να βρούμε μια συμβαστική λύση δηλαδή πριν από την Ολομέλεια. Αλλά και πάλι στη βάση της σημερινής ψηφοφορίας ε, θα ήθελα να συμμετάσχω σε άτυπες διαπραγματεύσεις και η απάντησή μου άρα είναι ναι. Ωραία λοιπόν. Ε, κάποιος από τους σκιώδεις που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Κύριος Βαντεκάμπ. Ωραία λοιπόν. Ο κύριος Μάντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχοντας ακούσει τις συζητήσεις πριν από τις ψηφοφορίες. Νομίζω ότι δεν θα ήταν φρόνιμο να στείλουμε μια ομάδα διαπραγμάτευσης στο όνομα αυτής της Επιτροπής και, στην στη συνέχεια να αλλάξουμε πορεία. Γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της, ε, όσον αφορά τη νομική γνωμάτευση. Άτυπα μπορούν βεβαίως να γίνουν πάντοτε διαπραγματεύσεις, αλλά όχι μια εντολή την οποία να μπορεί να διαπραγματευτεί η ομάδα αυτή για το κοινοβούλιο. Θα ήθελα να θέσω μία άλλη ερώτηση επί της διαδικασίας. Εγώ θεώρησα ότι θα γίνει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια και στη συνέχεια η κυρία Τσένοβα θα ζητήσει να μην γίνει η ψηφοφορία, να αναπευθεί στην Επιτροπή και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά θέματα εδώ. Αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσουμε να το πάμε στην Ολομέλεια σε δύο εβδομάδες. Ίσως θα μπορούσαμε να το αφήσουμε μέχρι την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ε, και στη συνέχεια να δούμε τι θα γίνει με την τολική ψηφοφορία. Ε, δεν ξέρω, θα ξεκινήσω διαπραγματεύσει την επόμενη εβδομάδα. Κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει ίσως θα ήταν καλό να περιμένουμε μέχρι την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ε, αλλιώς θα καθυστερήσει, θα μπορούσε να καθυστερήσει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Νομίζω θα πρέπει να πάρουμε τα πράγματα όπως έρθουν. Ε, και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Uh, Ωραία, λοιπόν, ας δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, δουλειά σας και, και για τις συμβαστικές τροπολογίες. Τώρα θα περάσουμε στην τροπολογία για την έκθεση του κυρίου Μάιερ. Θέλετε να πείτε κάτι πριν από την ψηφοφορία, κύριε Μάιερ. Όχι. Ωραία, λοιπόν. Τότε θα συνεχίσουμε αμέσως. Είσαστε έτοιμοι όλοι. Ωραία λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία Unblock υπαριθμό 1. Υπέρ του 1, unblock, κατά, απορρίπτεται. Θα έρθουμε στη συμβαστική τροπολογία 1, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα θα περάσουμε στα άρθρα, άρθρο 1. Τροπολογία 20 του εισηγητού, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 18 υπέρ. Α, ε, ήταν τμήμα του. Τότε το 21. Τροπολογία 21 του συγκητού υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Υπάρχουν αρκετέ ψηφοφορίε. Περάσουμε στη σημαντική τροπολογία περιφάνου 2 γιατί προηγουμένως κάποια άλλα καταπίπτουν. Δύο λοιπόν υπέρ κατά γκρίνεται. I think everything else Λοιπόν, όλα τα άλλα καταπίπτουν. 105 της κυρίας Ρούλε, υπέρ παρακαλώ, κατά απορρίπτεται. 1.57 από του υπέρ κατά εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά εγκρίνεται. 159. 159 είναι συμβατή με την 24. Θα τη βάλουμε σαν προσθήκη υπέρ 159 της κυρίας Ρούλε ως προσθήκη στην 24 του κυρίου Μάιερ. Υπέρ παρακαλώ, κατά, απορρίπτεται. 160. Α, και αυτή είναι συμβατή του κυρίου Γκάλ Πέλς. Υπέρ. Κατά. Αγκρίνεται. 21 καταπίπτει. 161 καταπίπτει. 162 υπέρ. Θα πρέπει να... 162 του κυρίου Κοφεράτη. Άρχεται η ψηφοφορία. πέραστες ψηφοφορίες Α, συγγνώμη. The τη closed. Πέρας της Απορρίπτεται. 21 ψήφοι κατά, 16 υπέρ. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν θα ψηφίσουμε την 163 του κυρίου Κάρας. Υπέρ. Κατά. Από... Απορρίπτεται. 164. Με μια προφορική τροπολογία. Έχει συμφωνηθεί προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 165. Υπέρ, κατά. Θα πρέπει να το ελέγξουμε. εγκρίθηκε 19 υπέρ 16 κατά. Η 166 καταπίπτει, 25 είχε αποσυρθεί, 22 καταπίπτει. Α, συγγνώμη, η 165 μπορεί να συμπεριληφθεί ως προσθήκη ότι είναι συμβατή. 166 υπέρ. Κατά. Α, γκρίνεται. 23 από την Επιτροπή Μεταφορών υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 167 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Υπέρ, συγγνώμη. Κατά. Εγκρίνεται. 168 είναι συμβατή. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 26, 26 έχει αποσυρθεί, 27 έχει αποσυρθεί, 24 των μεταφορών υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 25 της Επιτροπής Μεταφορών υπέρ, υπέρ της 25, κατά, απορρίπτεται, 169 της κυρίας Μακλάκρικιν υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 170, 170 καταπίπτει και 26. Η 28 του κυρίου Μάιερ με χωριστή ψηφοφορία. Ή μάλλον κατά τμήματα. Ε, τμήμα 1 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 27 το μεταφορών υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. 4 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. 198 μαζί με την 199 συνδέονται μεταξύ τους. Περ κατά απορρίπτεται και οι δύο απορρίπτονται. 200 υπέρ κατά επίσης απορρίπτεται. 200 υπέρ κατά εγκρίνεται. 202 προσθήκη υπέρ κατά απορρίπτεται. 203 υπέρ κατά απορρίπτεται. 204 υπέρ κατά απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά εγκρίνεται. 205 και 206 όχι έχει αποσυρθεί. 205 υπέρ κατά απορρίπτεται. 35 και 36 των μεταφορών υπέρ. Κατά εγκρίνεται. σημαντική τροπολογία 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 211 υπέρ κατά απορρίπτεται 212 υπέρ κατά εγκρίνεται 36 υπέρ κατά εγκρίνεται 213 προσθήκη υπέρ κατά απορρίπτεται 30, η τελευταία έχει αποσυρθεί 214 215 υπέρ κατά υπέρ 215 κατά εγκρίνεται μεταφορές 37 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική αεροπλογία 9 υπέρ κατά εγκρίνεται 38 υπέρ κατά εγκρίνεται 218 προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται μεταφορές 38 υπέρ όχι καταπίπτει 39 υπέρ κατά απορρίπτεται τραν 40 υπέρ κατά απορρίπτεται 219 υπέρ κατά εγκρίνεται 41 από την Επιτροπή Μεταφορών υπέρ. Θα πρέπει να επαληθεύσουμε. 41 από την Επιτροπή Μεταφορών. Άρχεται η ψηφοφορία. Κατά τμήματα. Α, όχι. 19 ε, υπέρ, 17 κατά εγκρίνεται. Η 39 καταπίπτει. Τροπολογία 40 υπέρ. Υπέρ τη 40. Κατά εγκρίνεται. Τη Επιτροπή Μεταφορών 42 ω προσθήκη. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 220 κατά τμήματα. Τμήμα 1. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 43 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. 221 ως προσθήκη υπέρ κατά απορρίπτεται από την Επιτροπή Μεταφορών του 44 ως προσθήκη. Υπέρ κατά όχι συγγνώμη υπέρ κατά Απορρίπτεται. 224 υπέρ. 222 ε, ε, συγγνώμη υπέρ. 225 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά εγκρίνεται. Και τέσσερις μαζί, ή ε, μάλλον όχι, 43 υπέρ κατά Ας επαληθέψουμε. Νομίζω ότι γκρίνεται, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται με δύο ψήφους. «47 από την Επιτροπή Μεταφορών υπέρ κατά απορρίπτεται». 44 του κυρίου Μάιερ υπέρ κατά εγκρίνεται 226 κατά πίπτη συμβαστική τροπολογία παριθμών 6 υπέρ κατά εγκρίνεται 48 από την Επιτροπή Μεταφορών υπέρ κατά απορρίπτεται 49 υπέρ κατά απορρίπτεται 230 υπέρ κατά Απορρίπτεται επίσης 231 υπέρ κατά. Εγκρίνεται 232 υπέρ κατά. Απορρίπτεται 233 υπέρ κατά. Απορρίπτεται επίσης 50 τραν υπέρ κατά επίσης απορρίπτεται 234 υπέρ κατά απορρίπτεται 235 υπέρ κατά εγκρίνεται 236 υπέρ κατά εγκρίνεται στραπλογία 7 υπέρ Α, ε, κατά τμήματα η 7 πρώτο τμήμα υπέρ Α γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση για τη συμβαστική τροπολογία 7, το πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Είναι μόνο μία λέξη. Ωραία, λοιπόν, θα ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Σαφώς. 237. Γιατί κατέπεσε η συμβαστική ρομολογία. Θα πάμε στο 241 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 242 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 246. Α, όχι, συγγνώμη. 46 είναι συμβατός προσθήκη υπέρ. Κατά εγκρίνεται 243. Δεν θα το ψηφίσουμε. 244 ως προσθήκη υπέρ. Κατά απορρίπτεται η 52 κατά πίπτη 245 υπέρ κατά απορρίπτεται 47 uh, sorry, 47, those in 47 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Μεταφορές 53 προσθήκη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 246 υπέρ. Η κατά εγκρίνεται. 247 και από την Επιτροπή Μεταφορών η 54 46. Should we vote on it anyway? We can sort it out later. Let's vote on. Let's vote on 247 and tram. 247 και 54 από την Επιτροπή Μεταφορών υπέρ και 247 κατά τι κάνει φιλελεύθερη. Είστε υπέρ. Κάνουμε διπλή επαλήθευση υπέρ. Κατά γκρίνεται. 249 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 55 από την Επιτροπή Μεταφορών υπέρ. Κατά. Επίσης απορρίπτεται. 250 υπέρ. Κατά. Ωραία, σε παληθεύσουμε. Για την 250 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες απορρίπτεται. 252 πέρ. Κατά εγκρίνεται. Δια... Συμβασική τροπολογία 8α υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 259 οφεράτη υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 έχει καταπέσει. 50 Το εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 ως προσθήκη. Με αυτές τις λέξεις που βλέπετε εδώ, υπέρ κατά εγκρίνεται. 2.60 με προφορική τροπολογία όπως βλέπετε εδώ ποιοι είναι υπέρ, κατά απορρίπτεται Τραν 60. Υπέρ. Υπέρ, παρακαλώ. Νομίζω πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τραν 60. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 47, ε, 17 υπέρ, 20 κατά. ένα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Εκείνο σε όλες καταπίπτουν. Πάμε στη τράν 62. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 51 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 263-264 καταπίπτουν. Α, είναι συμβατές. Υπέ... Η 265 είναι συμβατή επίσης. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 266 ε, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 267 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 268 και τραν 63. Είναι συμβατή. Τραν 63 ως προσθήκη. Τραν 63 ως προσθήκη υπέρ κατά απορρίπτεται. Τραν 64 υπέρ υπέρ κατά εγκρίνεται. 269 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τραν 65 το αντίστοιχο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά εγκρίνεται. Και πάμε στην τραν 65, το αντίστοιχο τμήμα, ως προσθήκη. Υπέρ. Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ε, μπορείτε να ψηφίσετε. Άρθρο 8. Μπορείτε να συντομεύετε λίγο. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στην τραν 69. Άρθρο 10 παράγραφος 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 302 καταπίπτει, η 301 είναι συμβατή, Α, καταπίπτει και αυτή. 62 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 306 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 303 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 304 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 370 70 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά εγκρίνεται 305 καταπίπτει 308 και 371 υπέρ ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά νομίζω πως καταπίπτουν, αλλά για να είμαστε σίγουροι Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 18 υπέρ, 17 κατά. Τώρα θέλω να ε, προχωράμε στην τραν 72. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τραν 73. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 64. Υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. Οπότε οι τρεις υπόλοιπες, 309, 10 και 11 καταπίπτουν, 374 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 313 είναι συμβατή, υπέρ, κατά, απορρίπτεται.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 Πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα για τη συμβαστική 11 που είναι λίγο παρακάτω στον κατάλογο ψηφοφορία. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ τη συμβαστική 11. Κατά εγκρίνεται. Οπότε τώρα πάμε πίσω. Γιατί όλα αυτά καταπίπτουν και πού πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Vote on Right? 319. Uh, those in... 319. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Uh, so we now go to 323. 323 τώρα. 323. Υπέρ. Α, όχι, έχει εξαταπέσει. Sorry, that, uh, 319 was adopted. Sorry, Sergio Cofferati. Α, συγγνώμη, κύριε Κοφεράτη. Πάμε στην τραν 78. Άρθρο 11, παράγραφος 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 327. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Yeah, if you can vote quickly, that's it, please. Um, rejected. Απορρίπτεται. 327 υπέρ κατά εγκρίνεται 67 Το εισηγητή με την προφορική υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά εγκρίνεται και πάμε στην 69 του εισηγητή υπέρ υπέρα παρακαλώ Uh, let's open the vote on this. Ηλεκτρονική. I think it's rejected, but we'll see. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται λοιπόν και περνάμε στην 341. Μακλάρκιν υπέρ... Και εδώ πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά νομίζω. 341 ψηφίζουμε.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 κατά εγκρίνεται. Τραν 81 συμβατή υπέρ κατά απορρίπτεται. 348 υπέρ κατά απορρίπτεται. 351 την ψηφίζουμε αυτήν. Μάλιστα.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 Μήπως μπορείτε να προχωρήσετε λίγο εσείς και να ελέγξετε. Απορρίπτεται 17 υπέρ 20 κατά. Και πάμε στην τραν 83, σωστά. Και το 353 υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 359 υπέρ, κατά απορρίπτεται. Πάμε στην 361. Okay. 361. Those υπέρ. Κατά. Καταπίπτει. 363. Ας το ψηφίσουμε έτσι κι αλλιώς. Το 63. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 364, 64, 365 και, και 84. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 366. 366 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 367 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 370 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 385 Κοφεράτη 371 ποιοι είναι υπέρ κατά απορρίπτονται 372 υπέρ κατά εγκρίνεται 73 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται 375 και 76 μαζί υπέρ κατά εγκρίνονται 74 και οι 377 καταπίπτουν 378 υπέρ κατά απορρίπτονται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβαστική 14 υπέρ κατά εγκρίνεται Πάμε στην τραν 89. Το αντίστοιχο τιμήμα Ποιοι είναι υπέρ. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τραν 89. Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is closed. Uh, that's rejected. Απορρίπτεται. 393 ε, υπέρ. Κατά απορρίπτεται 394 υπέρ κατά απορρίπτεται to 397 so we now have a block vote τώρα θα ψηφίσουμε unblock είναι η unblock ψηφοφορία 5 υπερθμών 5 ποιοι είναι υπέρ κατά απορρίπτεται Πάμε στην 399. Υπέρ κατά ε, απορρίπτεται. Transport 91. Υπέρ κατά εγκρίνεται. So do we not put So we now go to 79. Πάμε στην 79 του εισηγητή. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 412 υπέρ κατά απορρίπτεται 413 υπέρ κατά απορρίπτεται 80 έχει αποσύρθει 415 βερνιό με προφορική που έχετε εδώ υπέρ κατά εγκρίνεται 414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 εδώ έχουμε διάφορε της επιτροπή Μεταφορών. Μπορούμε να τι ψηφίσουμε μπλοκ. Πολύ ωραία. Transport 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 και 104. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται όλες. 418 και 105. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά εγκρίνονται. 419 υπέρ κατά εγκρίνεται. 420 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τραν και 107 υπέρ κατά απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 308 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τραν 109 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τραν 110 ως προσθήκη υπέρ κατά απορρίπτεται. 422 υπέρ κατά απορρίπτεται 423 υπέρ κατά απορρίπτεται 428 υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 424 υπέρ. Ε, <coughs> κατά. Εγκρίνεται. 426 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 427 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται τράνε 111 υπέρ. Α, καταπίπτει. Πάμε στην 430 τώρα, 430 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 431 καταπίπτει, 433, ποιοι είναι υπέρ, κατά, ε, ξανά παρακαλώ, 430 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 485 η 85 υπέρ κατά εγκρίνεται 435 υπέρ κατά εγκρίνεται 87 υπέρ κατά εγκρίνεται και πάμε στις αιτιολογικές σκέψη, συμβαστική 1 υπέρ α το έχουμε ψηφίσει μάλιστα Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 91 Έχει καταπέσει. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 92 και 93 έχουν καταπέσει, 94 δεν ψηφίζουμε, τραν 2 καταπίπτει, πάμε στην 95, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4, έχει ήδη ψηφιστεί. Και πάμε στην 99, 99 του εισηγητή. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 100, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά νομίζω ότι εγκρίνεται 101 Έλεγχος ηλεκτρονικός. Νομίζω πως εγκρίνεται. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σωστά τα έκρινα, αλλά καλό ήταν που το ελέγξαμε κιόλας. 103 υπέρ. Κατά. Αγκρίνεται. 102 καταπίπτει. 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 7 Το εισηγητή ως προσθήκη στη συμβιβαστική. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 9 του εισηγητή. Υπέρ, Υπέρ παρακαλώ. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 9. Τροπολογία 9. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20 προς 17. Τροπολογία 118 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική όχι 10 και του κυρίου Μάγερ υπέρ κατά εγκρίνεται Εκατόν είκοσι και τρανσπορτ 9 υπέρ κατά εγκρίνονται η 12 έχει καταπέσει 122 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται Οπότε καταπίπτει και 125. Η 130 είναι συμβατή. Α, η, 13 με συγχωρείτε, υπέρ. Υπέρ της 13. Ε, κατά εγκρίνεται. 123 είναι και αυτή συμβατή. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά στην 123. And that's rejected by two votes. 17 in favor, 9. Ε, ωραία, λοιπόν, ε, κατα, καταπίπτει αυτή. Πάμε στην 126 της κυρίας Στάιλερ. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 14 με προφορική. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 127 Κοφεράτη. Το αντίστοιχο τμήμα υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 127, 128, όλες αυτές καταπίπτουν. Και πάμε στην 15 του εισηγητή, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. «131 και 132 είναι ταυτόσιμες, υπέρ, Against. Those are carried. Κατά ε, εγκρίνονται. 134 υπέρ. Κατά. πρέπει να ψηφίσουμε κατά τμήματα το, το, 133 όχι, πέρασα στη 17 του εισηγητή. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 135 και 136 υπέρ, κατά. Εγκρίνονται. 18 ως προσθήκη υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 315 ως προσθήκη με αυτά τις λέξεις υπέρ, κατά απορρίπτεται 141 υπέρ κατά απορρίπτεται 316 υπέρ κατά απορρίπτεται Συμβιβαστική 8β με χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα. Τμήμα 1 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ, κατά Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Τρανο 17 υπέρ κατά απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης. Ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ.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 Λοιπόν, όσοι ήλθατε μόνο για να ψηφίσετε, παρακαλώ να καταλήψετε εισήγω στην αίθουσα, γιατί έχουμε άλλο ένα θέμα να συζητήσουμε σε για διάταξη. Κύριε Βίντεν Χόλτσερ, Βάιντεν Χόλτσερ, σε ένα λεπτό θα είμαστε έτοιμοι. Ένα λεπτάκι για να αποχωρήσουν όσοι δεν θέλουν να παραμείνουν στην αίθουσα. Πάρτε και τις κάρτες ψηφοφορίας μαζί σας. Γιατί βλέπω ότι πάνε και τις μαζεύουν ήδη από